Morning. Καλημέρα σας λέει ο Πρόεδρος. Good morning. Bonjour. Buenos días. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, καθίστε παρακαλώ. και να αρχίσουμε την συνεδρίαση της Επιτροπής των Πολιτικών Ελευθεριών και πρώτα πρώτα να εγκρίνουμε την ημερησία διάταξη. Έχω να σας πω επίσης ότι το σημείο για το δίκτυο συναγερμού και πληροφόρησης για τις κρίσιμες υποδομές, το σημείο 6, αναβλήθηκε προς συζήτηση σε άλλη συνάντηση. Παρακάτω, η συνάντηση των ε, συντονιστών και κλεισμένων, όπως πάντα, θα λάβει χώρα από τις 11.30 ε, μέχρι τις 12.30. Έχετε καμία ένσταση. Πάμε τώρα στις ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Πρώτον, όπως θα γνωρίζετε, μια αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας πήγε στην Ουάσιγκτον την περασμένη εβδομάδα. Συνάντησε μέλη του Κογκρέσου και της Αμερικανικής Κυβέρνησης. Και ενημερωθήκαμε ότι ήταν πάρα πολύ παραγωγικές και χρήσιμες για το μέλλον αυτές οι συναντήσεις. Όσον αφορά τα, τις πληροφορίες, τα δεδομένα που αφορούν τους επιβάτες αεροπόρων εταιριών και οπότε η έκθεση σχετική με αυτή την αποστολή πρόκειται να εγκριθεί την επόμενη φορά που θα συντηθούν οι συντονιστές. Όχι σήμερα, την επομένη φορά. Όταν ολοκληρωθεί η έκθεση. Τι θέλετε κύριε μου. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να πω όσο και να τώρα αναλώνω την, τον χρόνο της συνεδρίασης στα αγγλικά. Χαίρομαι, χαίρομαι που σας βλέπουμε. Yes. Tack. Ε, jag är lite besviken. Ξαναρχίζει. Όπως προανέφερα, με απογοήτευσε το ότι αρχίζουμε με τόση καθυστέρηση τις συνεδριάσεις μας. Είναι πάρα πολύ σημαντική η Επιτροπή μας διεξέρχεται τόσο σημαντικά ζητήματα και ποτέ, ποτέ δεν αρχίζουμε στην ώρα μας. Έχουμε τόσα θέματα να συζητήσουμε στην ημερησία διάταξη και αρχίσαμε στις 9 και 4. Θα μπορούσατε να στείλετε κάποια mail, να γράψετε κάτι, ούτω ώστε να τηρούμε το χρονοδιάγραμμα, γιατί υπάρχουν τόσο σημαντικά θέματα τα οποία πετούν χρόνο για να τα συναντήσουμε. Ελπίζω στο μέλλον να μπορούμε να αρχίσουμε στην ώρα μας. Βεβαίω, βεβαίω. Μα ήμασταν εδώ στι 9 και ε, πέρασαν λίγα λεφτάκια. Ε, είχα να πω κάτι σε κάποιου αδέλφου στην ε, αίθουσα. Φυσικά περίμενα ούτω ώστε να έρθουν όλοι και έχετε δίκιο, θα ληφθεί υπόψη αυτό το οποίο είπατε. Πρέπει να διεξέλθουμε όλα αυτά τα δύσκολα ζητήματα τη μέση διατάξεω και επομένω Επομένω, το αρχίσουμε στην ώρα μα είναι κάτι το οποίο πρέπει να το τηρεί η Επιτροπή μα. αυτό λαμβάνετε υπόψη αυτό το οποίο είπατε και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε τόσο ώστε να κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει, να κάνουμε ό,τι λέμε στη διάταξη, να αρχίζουμε στην ώρα μα. Ετησία, έκθεση όσον αφορά την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα των σημείων υπαριθμών 3. Είναι το πρώτο σημείο το οποίο θα συζητήσουμε και αφορά αυτήν την ετησία έκθεση. Έχουμε εδώ κάποιε διαδικαστικέ διατάξει όσον αφορά την πρόσβαση στο κοινό. Έχει αναλάβει την έκθεση η κυρία Χαουτάλα. Και θα εξετάσουμε τι πρακτικέ λεπτομέρειε σε σχέση με τα όσα προβλέπει ο κανονισμός του 1049 του 2001 όσον αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα. Και αυτό είναι κάπω πρόδρομη ρύθμιση του τι πρόκειται να ρυθμιστεί στο μέλλον, γιατί έχουμε και μια έκθεση που αφορά τον ίδιο κανονισμό που έχει αναλάβει ο, ο κύριος Κάσμαν. Και ουσιαστικά θα γίνει αναθεώρηση του 1049 και το 2008 μετά τη συνθήκη της Λισαβόνα, προέβη σε κάποια προπαρασκευή αυτής της ρύθμισης της Κομισιόν και τον Μάρτιο φέτος επίσης είχε κάποια πρόταση τροποποιητική για τον κανονισμό ε, τον ίδιο κομμουνισμό, τον 1049, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε έτσι έχει παραταθεί η ισχύς για να καλύψει όλα τα θεσμικά όργανα και τις υπηρεσίες κοινότητας. Ε, επίσης ε, είχαμε μία ακρόαση όσον αφορά την διαφάνεια. Το κάναμε εδώ, ήταν η κυρία Χαουτάλα, ο κύριος Κάσμαν, ο κύριος Γιατεμάκη. Επίσης συμμετέσχε από την ΑΦΚΟ, τη συνταγματική μας επιτροπή και τώρα δώσουμε το λόγο στην εισηγητριά μας την κυρία Χαουτάλα για να μας μιλήσει όσον αφορά αυτή την ε, έκθεση για την εφαρμογή του κανονισμού 1049 κάθετος 2001. Κυρία Χαουτάλα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Την περασμένη εβδομάδα η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών διοργάνωσε με επιτυχία αυτήν την ακρόαση όσον αφορά το πώς έχουν τα πράγματα για την πρόσβαση του κοινού και ε, με βοήθησε η κυρία Γιατεμάκη και ο κύριος Κάσμαν και εγώ ήμουν συνδιοργανώτρια και έτσι προέκυψε μια ξεκάθαρη εικόνα του τοπίου οπότε και παρά το γεγονός ότι το κανονιστικό ρυθμιστικό πλαίσιο είναι καταρχήν πάρα πολύ θετικό, δηλαδή ο κανονισμός 1049, ο οποίος ε, ε, ισχύει επί μία δεκαετία. Παρόλα αυτά διστάζουν τα θεσμικά όργανα για να κάνουν αυτό που πρέπει όσον αφορά του πολίτε και παρά τη θέση ισχύ τη Εθνική Λισαβόνα που προβλέπει και θεσπίζει ω θεμελιώδη δικαίωμα την πρόσβαση στα έγγραφα. Είναι θεμελιώδη δικαίωμα για να μπορούν να εμπλακούν και οι πολίτε στο γίγνεσθε. Και επομένω θεωρείται αυτό ότι είναι θεμέλιο οποιασδήποτε δημοκρατία. Εγώ έκανα το εξή. Εμελέτησα στην πράξη τι κάνουν τα θεσμικά όργανα για να εφαρμόσουν τον 1049 όσον αφορά τους πολίτες οι οποίοι ζητούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα έγγραφα. Πολύ συχνά μας λένε τα θεσμικά όργανα ότι ε, καλύψαμε τόσα αιτήματα, η κατάσταση είναι πάρα πολύ θετική, όμως δεν διαπιστώνουν ότι το πρόβλημα έγκυται στις υπόλοιπε περιπτώσεις. Δηλαδή εκεί που τα θεσμικά όργανα αρνούνται την πρόσβαση και πολλές φορές επικαλούνται ή καταχρώνται των ε, διατάξεων που προβλέπουν τις εξαιρέσει από τη δυνατότητα πρόσβασης όπου την προβλέπει ο 1049 επίσης σας υπενθυμίζω ότι ο κύριος Κάσμαν τώρα ε, ασχολείται με την έκθεση που αφορά την αναθεώρηση του σχετικού κανονισμού και πάρα πολύ σύντομα θα αποφασίσει η Επιτροπή μας τι θα κάνει, πώς θα αντιδράσει στη δεύτερη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκείνη η οποία ακολούθησε την πρώτη πρόταση δύο χρόνια αργότερα. Ούτως ώστε να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού σε σχέση με τα όσο επιτάσσει η της Λισαβόνας για να καλύψει ο κανονισμός τις υπόλοιπε υπηρεσίες και όργανα πέραν των τριών βασικών. Πολύ ενδιαφέρουσα η κατάσταση, η περίπτωση, διότι Έχουμε μια σειρά θεσμικών ε, οργάνων και υπηρεσιών, όπως η υπηρεσία εξωτερικής δράσης, η υπηρεσία για τη διατροφή, η, υπηρεσία για τα φάρμακα, που τώρα καλούνται να τηρήσουν αυτή την υποχρέωση. Και επίσης, τις αμέσως προηγούμενες εβδομάδες διαπιστώσαμε και με τις ακροάσεις ότι δεν έχουν εξοικειωθεί το οι και θα πρέπει τόσο και αυτέ οι υπηρεσίε να τηρήσουν τα πρόβλημα για την πρόσβαση στα έγγραφα. Κάτι άλλο επίση πολύ βασικό. Τα θεσμικά όργανα προφασίζονται κάποιου είδους λόγους που τους κάνουν να καθυστερούν την παροχή των πληροφοριών, την πρόσβαση στα έγγραφα, οπότε με το που καθυστερούν πια χάνει το νόημα του το αίτημα πρόσβαση στα έγγραφα. Επομένω, επιβάλλεται να γίνεται ταχεία εκπαιδεύση και να σέβονται την ανάγκη των πολιτών για ενημέρωση. Επίση, ο διαμεσολαβητή επιτέλεσε πάρα πολύ σημαντικό έργο γιατί τόνισε το ότι χρειάζεται να υπάρχει διαφάνεια και πρόσβαση στα έγγραφα. Και είπε ότι χρειάζεται μια πιο δυναμική πολιτικοί και υποτίθεται θεσμικά όργανα αλλά και οι πολίτες πρέπει να αποφύγουν διαδικασίες περιτές και να υπάρχει άμεση πρόσβαση μέσω ειδικών ε, μητρών και αρχείων υπάρχει άμεση πρόσβαση στα έγγραφα επίσης το νομικό καθεστώς τώρα που αφορά την υπόθεση της πρόσβασης είναι αρκετά άρτιο Γιατί η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι πάρα πολύ προοδευτική. Πάρα πολύ αποτελεσματική όσον αφορά την ερμηνεία τη σχετική νομοθεσία. Επομένω τώρα έχουν περισσότερη διαφάνεια. Και πάντω υπάρχει κάποια ανησυχητική τάση βασικά από το Συμβούλιο αλλά και σε άλλα θεσμικά όργανα, διότι αυτοί εμένουν ότι οι εξαιρέσει που προβλέπονται στον κανονισμό ε, επιδέχονται ευρύτατη ερμηνεία, κάτι το οποίο όμως αντιβαίνει στο δικαίωμα πληροφόρησης των πολιτών. Και βασική πρόφαση που χρησιμοποιούν τα θεσμικά όργανα και νομίζω ότι κάπως το κάνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι κάτι το οποίο ισχύει εδώ και κάποια χρονάκια που ονομάζεται ε, χρόνος, διάστημα, περίσκεψης προβληματισμού του θεσμικού οργάνου δηλαδή. Κατά τον τρόπο διστάζουν, διστροπούν, δεν δίνουν αυτά τα έγγραφα τα οποία χρειάζονται ούτως ώστε να δοθούν τα έγγραφα και έτσι δεν μπορεί να συμμετάσχει ο πολίτης στην λήψη της απόφασης διότι όμως δικαιούται να ξέρει, δικαιούται να ξέρει τι γίνεται πριν ληφθεί η τελική απόφαση. Πριν ληφθεί η απόφαση και να γίνεται εν μια διαβούλευση, μια ζήμωση δημόσια. Έχουμε τώρα κάποιες ε, υποθέσεις που έχουν υπορθεί στο δικαστήριο, ακόμα ε, εκκρεμωδικούν. Άρα θα πρέπει να δούμε τι γίνεται όσον αφορά την νομοθεσία και θεώρησα ότι είναι τρομερό, φρικτό το πόσα κράτη-μέλη δεν θέλουν να δημοσιεύσουν τις νομοθετικές προτάσεις. Και πιο εντυπωσιακή υπόθεση αφορά την υπηρεσία που ονομάζεται μια υπηρεσία τέλο πάντων που αφορά τις πληροφορίες και αρνείται το Συμβούλιο να δημοσιεύσει την θέση της κάθε χώρας όσον αφορά την προβασιμότητα στα έγγραφα. Παράδοξο αυτό γιατί η υπηρεσία ασχολείται ακριβώς με τα έγγραφα που το κάνει αυτό και έχουμε κάποιε σημαντικέ αποφάσει του δικαστηρίου που ορίζουν ότι η πρόφαση αυτή είναι αβάσιμη ό,τι χρησιμοποιεί το Συμβούλιο. Που λένε δηλαδή ότι ενώ ακόμα η νομοθετική διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν μπορούν να ξέρουν οι πολίτε. Μα δεν γίνεται αυτό και, και ας λένε ότι τα κράτη δεν μπορούν να αλλάζουν τη θέση τους. Μα δεν είναι έτσι. Οι πολίτες κατανοούν ότι πρόκειται για μια συνεχώς διαμορφούμενη κατάσταση και έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν. Και άλλωστε φυσικά και καταλαβαίνουν ότι τα κράτη μπορούν να αλλάξουν τη θέση τους. Επομένως, δεν είναι ντροπή, δεν πειράζει το να δημοσιεύσουν την, την πρόοδο των εργασιών για το νομοθέτημα. Οπότε, από πηγές του Συμβουλίου ακούμε ότι υπάρχει μεγάλη δεστροπία να συμμορφωθούν με το Συμβούλιο, με το, το Δικαστήριο. Αυτό είναι παράδοξο επίση διότι η συνήθεια τη Αβώνα ορίζει πρέπει να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε όλα είναι και περισσότερο δισταγμό και δυστροπία από το Συμβούλιο. Επίση, σας τονίζω μια άλλη υπόθεση που αφορά ε, ε, και τον διαμεσολαβητή, ο οποίο είναι πλάκι πέρσι και αφορούσε τον οργανισμό φαρμάκων σε σχέση με κάποιες εμπιστευτικές πληροφορίες που χαρακτηρίστηκαν έτσι. Χαρακτηρίστηκαν εμπιστευτικές και αφορούσαν την σύσταση κάποιων φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας. Και ορίζει ο Δημοσιευτής ότι θα έπρεπε να έχει δώσει ο οργανισμός φαρμάκων αυτές τις πληροφορίες και ότι αυτές τις πληροφορίες δικαιούνται να τις ξέρουν οι πολίτες. Αυτή ήταν η σύσταση του διαμεσολαβητού. Θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο ε, ανεφεί στην ε, ακρόαση την ε, περασμένη εβδομάδα οι κανόνες κατηγοριοποίησης των εγγράφων και εδώ είναι πρόβλημα. Πρόκειται για εσωτερικέ διαδικασίες της κάθε υπηρεσίας, του κάθε θεσμικού οργάνου και εκτός από τον κύριο Κάσμα στην εκθεσή του, αλλά και άλλοι που έκαναν την έρευνα την περασμένη εβδομάδα είπαν ότι η κατηγοριοποίηση των εγγράφων θα πρέπει να αντιστοιχεί στην κείμενη νομοθεσία και όχι να διέπεται από κάποιες ε, διατάξεις διαδικαστικές ε, επικουρικές δευτερογενούς δικαίου. Έχει ασχοληθεί και ο κ. Κάσμαν με αυτό όσον αφορά αυτή τη ρύθμιση που είναι πάρα πολύ λογική. Τώρα, έχουν βρει έναν αποτελεσματικό τρόπο τόσο ώστε να ξεγλιστράνε τα θεσμικά όργανα από την υποχρέωση της διαφάνειας γιατί αναβαθμίζουν υπερβολικά τα έγγραφά τους. Λένε περιορισμένη πρόσβασης, εμπιστευτικά, τα χαρακτηρίζουν πάρα, πάρα πολλά έγγραφα. Αυτή η κατηγορία διαβάθμισης δεν προβλέπεται πουθενά. Άρα θα πρέπει να θεσπιστεί νομοθεσία άρτια, σωστή. Και οι συνομοθέτε, οι βασικοί δηλαδή κοινοβούλιο και συμβούλιο, να αποφασίσουν ποιο είναι ο πιο αποτελεσματικό τρόπο, ώστε τα έγγραφα να χαρακτηρίζονται όπω πρέπει. Απόρριτα, άκρο απόρριτα, οτιδήποτε. Και να σταματήσει η κατηγοριοποίηση και ο χαρακτηρισμό των εγγράφων αποτελεί πρόφαση για την μη προσβασιμότητα. Ελπίζω ότι το έγγραφό μου θα σας δώσει κάποιες ιδέες ενδιαφέρουσε ε, χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα και πρόκειται να συντάξω αυτήν την ε, έκθεση σύντομα και ελπίζω ότι θα τα πούμε με τους και ηγητές επίσης σύντομα και τους ευχαριστώ όλους τους ε, συνεισηγητές και όδησηγητές, όλους γιατί δουλέψαμε σαν ομάδα πολύ αποτελεσματικά και επίσης σύντομα θα έχουμε στα χέρια μας και την έκθεση Κάσμα. Ε, Έχει πολύ, πολύ πράγμα. Ευχαριστώ. Κύριε Κάσμα, νομίζω ότι είστε πρώτος. <clears throat> Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Χάουταλα για την εξαιρετική παρουσίαση της ε, καταστάσεως της έκθεσής της. Βέβαια ουσιαστικά πρέπει, ε, αναφερόμαστε στην ε, πρακτική δηλαδή το πόσο λειτουργεί ο κανονισμός 1049 προτού να ισχύσει ο θεσμός. Οπότε πρέπει να δούμε αν υπάρχουν επαναλήψεις ή δυσκολία να διατεθούν δια διάφορα κείμενα διότι ουσιαστικά υπάρχει ε, ε, πλήρης ε, αρμονία μεταξύ του τι κάνει η κυρία ε, Χαουτάλα και τι κάνω εγώ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού 1049 διότι μιλάμε για την υπερβολική ταξινόμηση για να ξέρετε ότι ο κανονισμός 1049 βασίζεται στην πρόσβαση και συνήθως δεν υπάρχει άρνηση όταν υπάρχει άρνηση πρέπει να είναι αιτιολογημένη σύμφωνα με το άρθρο 4 των εξαιρέσεων ή το άρθρο 9 σχετικά με τα ευαίσθητα έγγραφα. Γι' αυτό και πολύ σωστά η κυρία Χαουτάλα ασχολείται με την ε, ταξινόμηση και με τα θέματα που και εγώ πραγματεύομαι. Ε, αν θέλουμε να είμαστε συνεκτικοί ε, όσον αφορά τη, ε, κάποιο έγγραφο το οποίο συνυπάρχει σε δύο θεσμικά όργανα και να έχουμε συνεκτική πρόσβαση πρέπει να έχουμε ένα ενιαίο σύνολο κανόνων όσο αναφορά το τα εγγραφά και εγώ βασίζομαι εις ε, το σύνολο των ε, κανονισμών όπως τους παρουσιάζει το Συμβούλιο διότι όταν υπάρχει μία ενιαία παρουσίαση πιστεύω ότι καταρχήν υπάρχει μία ενιαία πρόσβαση στα έγγραφα και είναι πιο εύκολο να έχει κανείς πρόσβαση στα έγγραφα αυτά. Η κυρία Χάουταλα αναφέρθηκε στην ακρόαση που είχαμε την περασμένη εβδομάδα ομάδα η οποία ήταν επιτυχής ιδίω για τους μη κυβερνητικού οργανισμούς ε, οι οποίοι έχουν πρόσβαση στα έγγραφα ή ορισμένοι στους οποίους αρνούνται να έχουν πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα διότι υπάρχουν οργανισμοί οι οποίοι έχουν επερβεί τα όρια όσον αφορά την ε, διαφάνεια και θεωρούν ότι ο κανονισμός το 1049 είναι μία βάση στην οποία πρέπει να ε, ε, βασίζεται ο εσωτερικός κανονισμός του οργανισμού τους και αυτό το βλέπουμε με διάφορα παραδείγματα όπως παραδείγματος χάρη την ετήσια έκθεση ε, του κανονισμού για την εφαρμογή του κανονισμού 1049 και έχουμε στην περίπτωση της βαβαρικής βίρας Λάγκερ μία ε, περίπτωση που βασίζεται σε μία ισορροπία μεταξύ συμφερόντων. Αφενός υπάρχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία αρνήθηκε την πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα διότι έλεγαν ότι θα υπήρχε παραβίαση ε, της προστασίας δεδομένων των ατόμων τα οποία περιλαμβάνονται σε αυτή την αγωγή και ε, δεν δόθηκαν αυτά τα έγγραφα στην περίπτωση Bavarian Lager αλλά πέραν αυτού πρέπει να υπάρχει και μια ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων δηλαδή δεν επαρκεί ε, το γεγονός ότι ορισμένοι αναφέρονται σε ένα έγγραφο να ε, μην επιτραπεί πρόσβαση ε, εις τα έγγραφα και στα στοιχεία και γι' αυτό πρέπει η ισορροπία μας να είναι πάρα πολύ καλά υπολογισμένη και να σέβεται και το συμφέρον του κοινού. Και το άλλο ενδιαφέρον στοιχείο και λέω ότι είναι ενδιαφέρον ε, είναι ε, το, η απόφαση του δικαστηρίου ECJ ε, σε σχέση με την θέση του, του δικαστηρίου όσο προς την αναθεώρηση του κανονισμού 1049. Δηλαδή προσπαθούσαν να διαπιστώσουν αν τα κράτη-μέλη ήθελαν να αναθεωρήσουν τον κανονισμό 1049, ήταν υπέρ της διαφάνειας ή προωθούσαν την αναθεώρηση και ένα από τα επιχειρήματα τα οποία ελήφθη υπόψη είναι και είναι θαυμάσιο να το διαβάσετε είναι σαν ένα μυθιστόρημα είδους Κάφκα διότι ε, ο ε, νομικός εκπρόσωπος λέγει ότι ε, αν δεν δημοσιευτεί δεν εφαρμόζονται οι αρχές αυτές διότι τότε το κοινό μπορεί να πιέσει τον νομοθέτη να αλλάξει γνώμη και ενδέχεται οι πολίτες να πιέσουν ε, για μία διαφοροποίηση. Είναι λοιπόν μία δικαστική απόφαση η οποία νομικά είναι πολύ αστεία διότι πρέπει κανείς να γελάσει για το πόσο ε, εμφανίζονται αυτά τα έγγραφα γι' αυτό και είναι τόσο σημαντικά. Δηλαδή ας μην κοροϊδεύουμε. Ε, είναι μια πολύ δύσκολη εποχή όσον αφορά το εθνικό περιβάλλον σαν κράτη-μέλη και πρέπει να δούμε εάν τα χρήματα που δαπανούμε για την Ευρώπη όντως αξίζουν τον κόπο και ε, αν σωστά ασχολούμεθα με τα θέματα αυτά. Γιατί πάντοτε μας λέει η Ευρώπη τι θα γίνει στη Σουηδία στην Πορτογαλία, στην Ιρλανδία, στην Ισπανία και ούτω καθεξής. Άπαξ και έχετε πρόσβαση σε έγγραφα του Συμβουλίου μπορείτε να δείτε πώς οι υπουργοί και οι κυβερνήσεις μας συζητούν και ψηφίζουν διότι οι ψηφοφορίες αυτές είναι εν κρυπτό. Οπότε ε, τα θέματα ακόμη και στα εθνικά κοινοβούλια δεν συζητούνται, δεν γνωρίζουν οι εθνικοί βουλευτές τι συζήτησαν ή πώς ψήφισαν οι υπουργοί τους στα Συμβούλια Υπουργών. Άπαξ και αυτά ανοίξουν στον έλεγχο του κοινού των πολιτών. Δεν είναι κακό αυτό. Καλό είναι να υπάρχει αυτή η δυνατότητα διοράσεως διότι ενδέχεται να έχουν αλλάξει γνώμη, να έχουν φτάσει σε μια συμβιβαστική λύση, να έχουν ψηφίσει. Μετά γυρίσουν βέβαια οι υπουργοί ε, στο Westminster, στο Εθνικό Κοινοβούλιο και πρέπει να λογοδοτήσουν συζητήσουν για την απόφαση την οποία έλαβαν. Πράγμα το οποίο θα καθησυχάσει τους πολίτες ότι η Ευρώπη δεν επιβάλλει. Υπήρξε συμφωνία των υπουργών μας που είναι στην κυβέρνηση και αυτό ο εμπεγμός των ευρωπαϊκών θεσμών πρέπει να σταματήσει και ιδίω είναι εις βάρος των προασπιστών της Ευρώπης και αυτά τα οποία παραδείγματος χάρη στο Sunday Times δίνει πολλά όπλα εις ε, του ευρωσκεπτικιστές για διάφορα προγράμματα τα οποία ήταν ε, πολύ επιτυχή και η Ευρώπη είναι το πιο ε, επιτυχές πρόγραμμα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρέπει λοιπόν να δούμε πού πρέπει να τραβήξουμε τη γραμμή. Βέβαια πρέπει να εξετάσουμε πού υπάρχει έλλειψη διαφανείας και γι' αυτό βάσει του κανονισμού 1049 εάν δεν διατίθεται ένα έγγραφο πρέπει να αιτιολογηθεί, να υπάρχει μια ελελογισμένη γνωμοδότηση. Εξού και θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογήσουμε τους τα τρία θεσμικά όργανα και σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τον κανονισμό 1049 θα είχα να πω ότι η πρόταση άργησε δύο χρόνια και δεν είναι πλέον αναγκαία διότι ότι η ε, ε, η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως το, άρθρο 15 έχει μία ήδη δυναμική. Είτε βασιζόμαστε στο 1049 ή όχι, το άρθρο 15 παράγραφος 3 ιδίως που αναφέρεται στην εμπλοκή των πολιτών στη δημοκρατική διαδικασία θα υπάρχει πάντοτε όσο θα υπάρχει και η Λισαβόνα. Είναι λοιπόν μία πολύ καλή άσκηση που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά δεν είναι αναγκαία και νομίζω ότι απλώς είναι ε, ένα πρόσχημα ε, για να βρουν τα ε, ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα τρόπο να βελτιώσουν την πρόσβαση πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την πρόσβαση και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το σύστημα. Κύριε Πρόεδρε, όντως μακρηγόρησα αλλά όσο περισσότερο ανοίγουμε τα θεσμικά μας όργανα τόσο περισσότερο θα αντιληφθούν οι πολίτες τι καλή δουλειά γίνεται και πώς η Ευρώπη πολλές φορές θεωρείται πρόσχημα για τις εθνικές κυβερνήσεις για ε, να αποφύγουν να εφαρμόσουν κάτι που δεν είναι πολύ δημοφιλές διότι ε, αυτό είναι ενάντιο στα συμφέροντα των 27 κρατών μελών. Ευχαριστούμε κύριε Κάσμαν. Έχουμε λοιπόν τώρα τα μέλη που μπορούν να λάβουν το λόγο. Βλέπω ο κύριος Μπουζουτήλ επιθυμεί το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο σκιώδης εισηγητής ε, του ΕΛΚ επί του θέματος είναι συνάδελφός μου η κυρία Ρενάτε Ζώμα που δυστυχώς δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ ε, λαμβάνω το λόγο εξ ονόματός της. Καταρχήν ευχαριστώ πολύ την κυρία Χάουταλα για μια πολύ ενδιαφέρουσα εισήγηση και θα μου επιτρέψετε να εκφράσω τις απόψεις του ΕΛΚ απόψεις οι οποίες ε, κατά κάποιον τρόπο προσφέρουν μια διαφοροποιημένη προσέγγιση σε σχέση με αυτά τα οποία ανέφεραν οι προηγούμενοι ομιλητές. Πρώτα απ' όλα ε, ξεκινάω με το εξή σχόλιο. Για μας το σημείο κίνησης πράγματι είναι πως η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να γίνει περισσότερο κατανοητή και περισσότερο διαφανής προς τα έξω. Αυτό λοιπόν είναι ένα κέριο ερώτημα. Πώς μπορούμε να προσφέρουμε στους πολίτες τα έγγραφα που χρειάζονται για να κατανοήσουν καλύτερα τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το τι ακριβώς πράττουμε εδώ. Είναι λοιπόν απαραίτητο να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην, ε, στον ανοιχτή Ένωση και στο να είναι διαφανής αφενός και αφετέρου στην αποτελεσματικότητά της ε, ακούστηκαν ορισμένες απόψεις όπως ε, παραδείγματο χάρη ε, κοινό εικονικό χώρος που προσφέρεται και αναφέρεται στα έγγραφα κατά την άποψή μας αν συνέβαινε κάτι τέτοιο θα καταλήγαμε με μια πλημμυρίδα εγγράφων που δεν είναι απαραίτητο ότι όλα αυτά τα έγγραφα ε, ενδιαφέρουν το κοινό. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε και πολύ προσεκτικοί για το κατά πόσον όλα αυτά θα συμβάλλουν στη διαφάνεια ή μήπως ε, τελικά συμβάλλουν ε, στο να καταστραφεί και αυτός ο χώρος που χρειαζόμαστε στη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας. Οι προηγούμενοι μιλητές είπαν ότι οι ε, θέσεις του Συμβουλίου για τα έγγραφα που δημοσιεύει ή όχι ε, μοιάζουν σαν ε, βιβλίο του Κάφκα. Ίσως είναι αλήθεια ότι αν τελικά το Συμβούλιο ή ένα κράτος μέλος είναι αναγκασμένο να δημοσιεύει τη θέση του, τότε ενδέχεται το Συμβούλιο ή το κράτος μελού να δημοσιεύει κάτι που δεν λέει απολύτως τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να δούμε κατά πόσον αυτό θα συμβάλλει στη διαφάνεια ή αντίθετα μήπως την ε, αναχαιτήσει. Και εδώ υπάρχει ε, ένα επιχείρημα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, ότι δηλαδή το θέμα δεν πρέπει να απορρίπτεται ως ε, καυκικό, είναι ένα θεμελιωμένο επιχείρημα και πρέπει να το αντιμετωπίζουμε δεν πιστεύω ότι πρέπει να επιλέξουμε μια τέτοια προσέγγιση όπου να μην δημοσιεύεται κανένα έγγραφο του Συμβουλίου. Καθ' άλλο, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η διαδικασία της δημοσίευσης δεν θα πρέπει να λαμβάνει με τέτοιο τρόπο, χώρα με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να παρεμποδίζει τα κράτη-μέλη να εκφράζουν την πραγματική τους άποψη. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες ε, δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στην περίπτωση ορισμένων φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι οι οργανισμοί Europol και Frontex. Πράγματι πρόκειται για πολύ ευαίσθητες πληροφορίες που εμπλέκονται με αυτούς τους δύο φορείς. Δεν είναι εύκολο να δημοσιεύει κανείς τα πάντα προς ε, τα έξω, αλλά ε, πρέπει να υπάρχει σύνεση όταν πρόκειται για ευαίσθητα έγγραφα, κυρίως όσον αφορά αυτούς τους οργανισμούς που ασχολούνται με την εφαρμογή του νόμου. Ολοκληρώνοντας λοιπόν, θέλω να πω το εξή. Υπάρχουν τρία προβλήματα κατά την άποψή μας. Πρώτον, όσον αφορά τη συνεχιζόμενη σύγχυση ανάμεσα αφενός στην πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα και αφετέρου στη θεσμική πρόσβαση. Δηλαδή, με λίγα λόγια, στην πρόσβαση που έχουμε εμείς ως θεσμοί. Νομίζω λοιπόν ότι δεν πρέπει να μιλάμε ε, για αυτά τα δύο θέματα σαν ένα ακριβώ τα ίδια, γιατί αυτό δεν εξυπηρετεί την όλη συζήτηση. Κατόπιν, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα με τον ορισμό. Τον ορισμό εγγράφων που πολλές φορές συγχέεται με τον ορισμό της πληροφορία, τον ορισμό του θεσμού και τον ορισμό του νομοθέτη. Η ε, πληροφορία επίσης του ε, κυρίαρχου ή μεγάλου ενδιαφέροντος από πλευρά κοινού και αυτός ο ορισμός δεν υπάρχει. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί κυρίως όσον αφορά τον περιορισμό ε, ε, του προβληματισμού, της σκέψης. Εμείς ως νομοθέτες θα πρέπει να είμαστε σε θέση να συζητάμε ε, με κάποια αξιοπιστία γιατί με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε πραγματικά να ε, ανταλλάξουμε απόψεις. Η πλήρης δημοσίευση των σκέψεών μας και των εγγράφων μας ενδέχεται να εμποδίσει εμάς τους ίδιους στο να εκφραστούμε ελεύθερα. Προφανώς βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο, δηλαδή το ΕΛΚ δεν διαφωνεί με αυτά που είπε η κυρία Χάουταλα, αλλά από την άλλη εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχει μια κατά τη διαφοροποιημένη προσέγγιση, λιγάκι διαφορετική αν θέλετε, μια προσέγγιση που και αυτή νομίζω θα πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Μπουζουτήλ. Ε, βλέπω τον κύριο Ντεγιόν που επιθυμεί να λάβει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, πρέπει να ευχαριστήσω τόσο την εισηγήτρια, την κυρία Χάουταλα, όσο και τον κύριο Κάσμαν. Διότι πρώτα απ' όλα μας προσέφεραν πλούσιο υλικό, το οποίο είναι πολύ χρήσιμο και ο Μάικλ σε σχέση με αυτά που είπε ήταν πολύ ενδιαφέροντα όταν αναφέρθηκε στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και εγώ θέλω να εστιάσω την προσοχή μου ακριβώς σε αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ στις Βρυξέλλες αλλά και στο Στρασβούργο τα καταφέρνουμε πάρα πολύ καλά το να αποκλείουμε τους πολίτες όταν τα πράγματα γίνονται ουσιαστικά ενδιαφέρονται για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας υποθέσουμε ότι εγώ είμαι πολίτης και διαβάζω μια εφημερίδα. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι το αποτέλεσμα που απορρέει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό εμένα δεν μου αρέσει και δεν άρεσε και στους Φιλανδούς από ό,τι είδατε γιατί έφτασαν σχεδόν το 20% οι ακροδεξιοί. Νομίζω λοιπόν ότι αξίζει το να ακούσουμε την άποψη των πολιτών και εμείς ως κόμμα προσπαθούμε λιγάκι και να αναζωογονήσουμε τη συζήτηση στη δική μου τη χώρα για το τι ακριβώς συμβαίνει με την οικονομική διακυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή λαμβάνονται εξόχως ενδιαφέρουσες και αποφασιστικές αποφάσεις και πολύ λίγοι γνωρίζουν τι πραγματικά διαδραματίζεται. Εάν λοιπόν μπορούμε να ανοίξουμε προς τα έξω και ε, βλέποντας ότι το ένα κράτος ε, μέλος συγκρούεται με το άλλο, ότι υπάρχει ουσιαστικά ουσιαστική σύγκρουση συμφερόντων. Αυτό δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να φοβόμαστε. Ε, αυτό είναι κάτι που δημιουργεί ένταση. Όλοι οι πολίτες ενδιαφέρονται να γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Αυτές τις μέρες ε, πολλοί έχουν ε, ε, από την τηλεόραση γιατί βλέπουν διάφορα σοκ και ξαφνικά βλέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βλέπουν ένα κτίριο και κάποιο αναφέρει το αποτέλεσμα απλά μια συνδιάσκεψη. Αυτό είναι ε, βαρετό για τους πολίτες. Εκείνο που ενδιαφέρει είναι η τσακωμή ανάμεσα στα κράτη-μέλη και αν θέλετε και η τσακωμή ανάμεσα στα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή είναι λοιπόν η μόνη σύσταση που θέλω να κάνω ε, σε αυτά τα οποία είπε η κυρία Χάουτελ. Ας μην ξεχνάμε του εαυτού μας όταν τα πράγματα γίνονται ουσιαστικά ενδιαφέροντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε στον τριμερή διάλογο, εκεί κλείνουμε τι πόρτε και δεν αφήνουμε τίποτα να διαρρεύσει. Οι πολίτες όμως αυτό ακριβώ θέλουν να μάθουν. Αν λοιπόν τολμήσουμε να ανοίξουμε τις πόρτες και να πούμε ότι ξέρετε δεν μας ενδιαφέρει η απόφαση ή δεν μας αρέσει η απόφαση του Συμβουλίου ας πούμε για το άσυλο εμείς επιθυμούμε το Συμβούλιο να λάβει μια άλλη απόφαση τότε και οι πολίτες θα δουν ότι και βέβαια προβαίνουμε σε συμβασμούς αλλά είμαστε και εμείς καθοριστικό στοιχείο της δημοκρατίας και νομίζω ότι αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε κύριε Ντεγιόγκ. Εάν λοιπόν ε, δεν επιθυμεί κανείς άλλος ε, να λάβει το λόγο σε αυτή τη συζήτηση, θα επανέλθουμε στην κυρία Χάουταλα για τις ε, καταληκτικές της παρατηρήσεις. Πρόεδρε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Μπούσουτιλ που τώρα δεν με ακούει. Σάιμον είπα ότι σου είμαι ευγνώμων διότι διατύπωσες όλα επί των οποίων διαφωνείς γιατί νομίζω ότι θα πρέπει τελικά να συμφωνήσουμε στην Επιτροπή μας ίσως ε, και ε, στην συνάντηση των σκιωδών εισηγητών πρέπει να έρθεις και εσύ γιατί θα πρέπει να συνοηθούμε αλλιώς στο Κοινοβούλιο δεν θα μπορέσει να προωθήσει τις θέσεις του. Εδώ και χρόνια το διαπραγματευόμαστε. Να σας πω τώρα κάποιες ε, απλές απαντήσεις σε αυτό το οποίο ερώτησες και σημειώνω και πάλι ότι θα πρέπει όλα αυτά να ζητηθούν και θα πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Επομένως, αυτή η σύγχυση μεταξύ της πρόσβασης στα έγγραφα και της προνομιακής σχέσης πρόσβασης σε αυτά όσον αφορά το κοινοβούλιο είναι κάτι το οποίο αφορά και αυτά τα οποία έχουμε πει εμεί όσον αφορά τι διαμορφωτικέ εντολέ για τι διεθνεί συμφωνίε, ούτω ώστε τελικά να μπορέσουμε να δώσουμε το πράσινο φω για τι σχετικέ συμφωνίε. Όχι, όχι, όχι. Ελπίζω ότι δεν είναι αποκλειστικό κανένα μυστικό, αλλά νομίζω ότι η νομική μα υπηρεσία έχει γνωμοδοτήσει κατά τρόπο πάρα πολύ σωστό σε σχέση με το πόσο θα πρέπει το Κοινοβούλιο να έχει πρόσβαση ε, στη διαπαντευτική εντολή της Ένωσης για την ε, Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και γιατί το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει εκεί πέρα αυτή την πρόσβαση, διότι και εμείς έχουμε το δικαίωμα να γνωρίζουμε το τι είναι υποδιαπραγμάτευση για ένα θέμα στο οποίο εμείς τελικά θα πρέπει να δώσουμε ή να μην δώσουμε πράσινο φως. Και οι πολίτες θέλουν να γνωρίζουν, οπότε και εμείς θα πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ του δικαιώματος των πολιτών και του δικού μας δικαιώματος, γιατί υπάρχει κάποια σχέση. Σε ευχαριστώ που ανέφερες ε, ότι είναι προβληματικό αυτό το διάστημα διασκέψεως του Κοινοβουλίου, space to think. Θα πρέπει να υπάρξει ένα όριο, πέρα από το οποίο και διαβουλεύσεις κάποιου μικροργάνου θα πρέπει να δημοσιοποιούνται. Όχι. Όταν τον εισηγητή, ας πούμε, μια έκθεσης, ε, όταν κάνει τις επαφές του, τα σχετικά πρακτικά, δεν αποτελούν πρακτικά ψηφίσμαση επίσημε συνεδρίες, επομένως δεν υπάρχει εκεί υποχρέωση να δημοσιοποιούνται. Και επίσης όσον αφορά τους ορισμούς, το κατά πόσον ε, είναι δημοσίου συμφέροντος, τελικά θα κρίνει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και τα άλλα δικαστήρια της κοινότητας. Ε, δεν πάνε και κάθε μέρα οι πολίτες στα δικαστήρια αυτά για να κατοχήσουν τα δικαιώματά τους και τώρα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό αυτό το οποίο έκαναν οι, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες προσέφεραν στα δικαστήρια για να ε, γίνει η σωστή ερμηνεία του νόμου. Άρα όντως χρειάζεται να οριστούν καλύτερα αυτές οι διατάξεις, αυτοί οι ορισμοί που είναι αρκετά αόριστοι. Τώρα όσον αφορά ε, αυτό τον ιδιατό χώρο τον εικονικό αυτό χώρο που θα δημιουργήσει μια πλημμυρίδα εγγράφων τα είπε καλά και ο όλα τελικά το θέμα είναι ότι είναι δικαίωμα του πολίτη να ζητεί να πληροφορηθεί το πρόγραμμα των εγγράφων και δεν το αποφασίζει, δεν το κρίνει το θεσμικό όργανο επί δικαιωμάτων, επί ε, εγγράφων μπορεί να το κάνει αυτό. Να λοιπόν, που μπαίνει το θέμα του εικονικού χώρου. Άρα θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση σε σχέση με το τι μπορεί να δει ο πολίτης. Βέβαια, σαφώς δεν είναι ενδιαφέροντα όλα τα έγγραφα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά έγγραφα τα οποία ποτέ δεν δημοσιοποιούνται γιατί δεν υπάρχει αυτός ο κοινό εικονικός χώρος. Άλλωστε υπάρχει ε, συνένεση μεταξύ του ΕΛΚ και των υπολείπων κομμάτων. Έτσι είναι η κατάσταση τελευταία διετία. Και μας κατηγορεί το Συμβουλίο ότι δεν συμπράττουμε για τη θέση νομοθεσίας. Επομένως, ας τα βρούμε και ας διευκρινίσουμε την κατάσταση. Κυρία Χάτουλα, σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα προχωρούμε στο επόμενο σημείο, το υπαριθμό 4 για την κινητικότητα των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε θα πρέπει να σας πω ότι στη συνέχεια θα έχουμε την συζήτηση ενός σχεδίου εκθέσεως που θα παρουσιάσει η κυρία Μπλίνκεβιτσιούτε αλλά θα κάνουμε και τη σχετική ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρα σας πενθυμίζω ότι θα πρέπει να έχετε την ε, κάρτα της ψηφοφορίας, να σας τη φέρουν τέλος πάντων, αν δεν την έχετε. Επομένως, πάμε στο σημείο παριθμών 4. Για να ακούσουμε την εισήγηση της κυρίας Μπλίνκεβιτσιούτε όσον αφορά το σχέδιο της έκθεσης για την προώθηση της κινητικότητας των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρίως αρμόδια επιτροπή είναι η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης και εκεί η συγκητή είναι ο κύριος Γιούρου Γεράνου, συγγνώμη, Ουγγουράνου, διορθώνει ο πρόεδρος. Όμως, πρώτα-πρώτα, να μας πει δυο λόγια η συγκήτρια, η κυρία Σιούντε. Και κατόπιν ακούσουμε τι γίνεται με, τη, με την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατόπιν θα συζητήσουμε. Μπλίνκεβιτσιούτε. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πιστεύω ότι η έκθεση του κυρίου Ουγγουριάνου βασίζεται στα μέτρα τα οποία θα προωθήσουν την κινητικότητα των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα καταλύσουν τα εμπόδια και ε, θα διευκολύνουν την κινητικότητα των εργαζομένων. Πιστεύω επίσης ότι είναι βασικό να τονίσουμε στην έκθεση αυτή τη σημασία της προστασίας των δικαιωμάτων των μετακινουμένων εργαζομένων ε, και να υπάρχει δυνατότητα αποκατάστασης, ε, να υπάρχουν δηλαδή ε, και αποτελεσματικές κυρώσεις και δυνατότητες διορθώσεως αποκατάστασης, της αποζημίωσης εφόσον, και, εφόσον έχουν πληγεί τα δικαιώματα των εργαζομένων αυτών. Προσπαθώ επίσης να αναφέρω αναφερθώ εις ε, τη σημασία των αμέσων και μέσων διακρίσεων εις βάρος των εργαζομένων ή ε, της ε, κατάχρησης της ε, ε, θέσεως ορισμένων. Δηλαδή ε, πολλές φορές οι εργαζόμενοι δεν καταλαβαίνουν τη γλώσσα, δεν γνωρίζουν ότι εθνικές νομικές διατάξεις και μειονεκτούν. Γι' αυτό και θα πρέπει να υπάρξει εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με τις ελάχιστες πληροφορίες που ο εργοδότης πρέπει να προσφέρει στον εργαζόμενο και ε, στη σχέση που βασίζεται στη σύμβαση εργασίας. Δηλαδή θα πρέπει να ξέρει πού εδρεύει ο εργοδότης ε, και ο εργαζόμενος, πόσες ώρες θα εργάζεται, τι διάστημα θα καλύπτει η σύμβαση ε, χρονικά και θα πρέπει να υπάρξουν εκτενείς ε, πληροφορίες που θα διετίθενται στον εργαζόμενο σχετικά με την απασχόλησή του Επιπλέον δε νομίζω ότι πρέπει να ε, καταπολεμήσουμε την κατάχρηση της, ε, των δικαιωμάτων των ε, εργαζομένων. Πέραν αυτού, οι εργαζόμενοι πρέπει να ελέγχουν ε, αν εφαρμόζονται σωστά οι διάφορες διατάξεις, να γνωρίζουμε πώς λειτουργούν τα γραφεία ευρέσεως εργασίας και τονίζω επιπλέον ότι ε, υπάρχουν και κοινωνικοί παράγοντες που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία πέραν των επαγγελματικών οργανώσεων οργανώσεων. Γι' αυτό και αυτό θα είναι πολύ σημαντικό για να αποφύγουμε οποιαδήποτε κατάχρηση των δικαιωμάτων των μετακινούμενων εργαζομένων και η γνώμη μου, η γνωμοδότησή μου καταρχήν ήταν πιο εκτενής αλλά χρειάστηκε να την να μειώσω την έκτασή της και ε, γι' αυτό μπορείτε να προτείνετε τροπολογίες σχετικά με τα μέλη της οικογενείας των εργαζομένων ή στις συνθήκες εργασίας τους. προσλέπω ή στις παρατηρήσεις σας και τροπολογίες σας και τα σχόλιά σας. Ελπίζω ότι θα έχουμε μία εποφελή συζήτηση, θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε το κείμενο και να καταλήξουμε σε καλύτερη, ε, ε, ε, καλύτερη δυνατότητα. Κυρία Μπλινκεβιτσούτε, τώρα θα μιλήσει ο κύριος Κοντιζάς εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε συμφωνώ πλήρως με τις ανησυχίες τις οποίες εξέφρασε η εισηγήτρια σχετικά με την αποτελεσματικότητα του δικαίου και τα διάφορα θέματα τα οποία έθιξε η εισηγήτρια διότι όντως πρόκειται για ένα ουσιαστικό δικαίωμα το οποίο ισχύει από τη συνθήκη της Ρώμης δηλαδή η δυνατότητα ελεύθερης διακίνησης των εργαζομένων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει ένα πολύ ε, βασικό άρθρο της συνθήκης, υπάρχει ε, και ένας κανονισμός και μία οδηγία που αναφέρονται στο θέμα αυτό, αλλά βλέπουμε ότι συχνά οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν δυσκολία όταν ε, μετακινούνται, ιδίως όταν προέρχονται από τις νεοεισηγμένες χώρες για να επιβάλλουν τα δικαιώματά τους και την ε, ε, ισότητά σου με τους εθνικούς εργαζόμενους. Είναι θέμα πληροφόρησης και πέρυσι έγινε μια ουσιαστική πληροφόρηση ε, σχετικά με τους μετακινούμενους εργαζόμενους και υπάρχει και μια ανακοίνωση νομική η οποία προσπαθεί να παρουσιάσει το κοινοτικό και εκτιμένο επί του θέματος. Επίσης υπάρχει μία Συμβουλευτική Επιτροπή ε, για τα Δικαιώματα των Εργαζομένων όπου εκπροσωπούνται ε, όλοι οι ενδιαφερόμενοι και όπου συζητάμε τα θέματα και προσπαθούμε να ε, βρούμε λύσεις σε θέματα κοινοτικού δικαίου. Αλλά ουσιαστικά αυτό ούτως ή άλλως συνάδει και με το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κοιτάζουμε να αναθεωρήσουμε την νομοθεσία, να την καταστήσουμε πιο αποτελεσματική και ε, θέλουμε να αναθεωρήσουμε το κείμενο το κείμενο που αναφέρεται εις το θέμα αυτό κατά τρόπον ώστε ε, να γίνει πιο αποτελεσματικό και ε, κάνουμε μία πρωτοβουλία του χρόνου μάλλον και αυτή τη στιγμή προσπαθούμε ε, να ε, ε, κάνουμε μία αξιολόγηση επιπτώσεων σχετικά με το πόσο θα μπορέσουν να γίνουν πιο αποτελεσματικά αυτά τα θέματα και οι σχετικές διατάξεις και γι' αυτό και η έκθεση αυτής της Επιτροπής θα οδηγήσει προς την ίδια κατεύθυνση όσον αφορά τις συζητήσεις που θα γίνουν και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι πολύ πιο εύκολο να καταρτήσει τις αρμόδιες προτάσεις κατά τρόπον πιο αποτελεσματικό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κοντιζά και τώρα λοιπόν ξεκινάει η συζήτηση ε, με, τους, τα μέλη της Επιτροπής. Ο κύριος Γιακολίνο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή την έκθεση της συναδέλφου κυρίας Μπλίνκεβιτς και θέλω να σας πω ότι συμφωνώ με πάρα πολλά από αυτά τα οποία ανέφερε. Η έκθεσή της είναι πολύ συγκεκριμένη και είναι σωστό ότι τα κράτη-μέλη οφείλουν και αυτά να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, ε, να ε, μην υπάρχει εκμετάλλευση των εργαζομένων και να υπάρχει ένα σαφές νομικό πλαίσιο, ένα πλαίσιο για τη νόμιμη μετανάστευση. Αυτές είναι οι δύο οδηγίε ε, τις οποίες συζητάμε μαζί με τον συνάδελφο κύριο Μωράης αφενός ε, ε, πρόκειται για τους εποχιακούς εργαζόμενους και φετερού η έκθεση. Αυτό είναι σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Πρέπει λοιπόν να καλέσουμε τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν την αρχή της ελεγγύης για την αλήθεια ότι οι πολίτες ε, των τρίτων χωρών μπορούν πράγματι να βοηθήσουν με τις εισφορές τους έτσι ώστε να αυξηθεί η ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν πρέπει λοιπόν κυρίως τώρα, σε αυτή την ιδιαίτερη περίοδο που βιώνουμε, να ξεχνάμε την αρχή της αλληλεγγύης ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Η αρχή αυτή δυστυχώς πολλές φορές ε, παραβιάζεται. Και είμαι πεπισμένος ότι η γνωμοδότηση αυτή μπορεί να συμβάλλει σημαντικά ευρύτερα στο θέμα, ένα θέμα που συζητιέται και σε άλλες βέβαια επιτροπές και είμαι επίσης πεπισμένος κύριε Πρόεδρε ότι πρέπει να ενισχύσουμε ενισχύσουμε την αρχή της πραγματικής αλληλεγγύης που σήμερα με το άρθρο 80 περισσότερο από ποτέ πρέπει να αποτελεί τη βάση οποιασδήποτε μορφής διαλόγου και οποιασδήποτε επικοδομητικής προσέγγισης από τα άλλα ευρωπαϊκά όργανα ξεκινώντας από το Συμβούλιο. Ευχαριστούμε κύριε Γιακολίνο. Ο κύριος Κέρκοπ. Παρακαλώ. Πρόεδρε, απλά θέλω και εγώ να προσθέσω κάτι. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω θερμά την εισηγήτρια για τη δουλειά της και επίσης να πω ότι κατανοώ τη σχέση ανάμεσα σε αυτή την οδηγία και την προτινόμενη οδηγία για τους εποχιακούς εργαζόμενους. Ε, από την εμπειρία μου οι μετανάστες εργαζόμενοι μπορούν να είναι αντικείμενο κάκιστης εκμετάλλευσης ε, είτε είναι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε όχι. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίζουν τους ε, πολίτες αυτούς ε, με το σωστό τρόπο. Σαφώς και πρέπει να υπάρχει συνεργασία ανάμεσα σε αρμόδιες αρχές. Πρέπει όμως να εκφράσω και μία ανησυχία μου που έχει έμεσα σχέση με αυτή την έκθεση και γενικότερα με το θέμα της κινητικότητας των εργαζομένων. Όταν ένας εργαζόμενος έχει ειδική τεχνογνωσία νομίζω είναι πολύ σημαντικό ότι χρειαζόμαστε αυτούς τους εργαζόμενους και αυτοί πρέπει να έχουν και κάποια σχέση με τους εργοδότες τους. Ε, είχαμε μία πολύ σοβαρή περίπτωση όπου ένας γιατρός ήρθε στη Βρετανία από τη Γερμανία. Το ιστορικό του στη Γερμανία ήταν ότι ερχόταν από την Ιγυρία. Δεν, μόλουσε, μίλουσε καλά γερμανικά αλλά μιλούσε πολύ καλά αγγλικά και πέρασε μέσα από τις αρμόδιες αρχές ε, στη Μεγάλη Βρετανία μέσα από διάφορα κανάλια πέρασε το γλωσσικό στοιχείο, αλλά δεν είχε γνώσει ιατρική, δεν είχε επαρκή γνώση ιατρική. Ένα ασθενή μάλιστα πέθανε. Και γι' αυτό τον ξανάδιωξαν, τον έστειλαν πίσω στη Γερμανία. Οι Γερμανοί όμω εξακολουθούν να τον απασχολούν. Και τώρα είναι και 65 χρονών περίπου. Αυτό λοιπόν είναι μια πολύ σοβαρή περίπτωση. Σίγουρα και πρέπει να ε, στηρίζουμε την κινητικότητα, αλλά πρέπει να καλύπτονται και κάποιε προδιαγραφέ, αν δεν θέλουμε να δημιουργούμε κινδύνου για τους ε, πολίτες. Κατόπιν τούτου, βεβαίως και στηρίζω την έκθεση, είναι πάρα πολύ καλή, αλλά πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη, έχοντας ε, κατά νου ε, τους μετανάστες εργαζόμενους και το τι ακριβώς έχουν κάνει πριν τελικά αν θέλετε επιβαρύνουν ε, τα κράτη-μέλη τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις ε, αρνούνται την κινητικότητα αν δεν καλύπτονται ορισμένες προδιαγραφές, ορισμένοι όροι. Πρόεδρος. Δεν ακούω. Α, πρόεδρος. Η συγγήτρια, η κυρία Μπλίνκε για τις τελικές ε, παρατηρήσεις της, παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Λέει κύριε Μπλίνκεβιτσιούτε, σας ευχαριστώ πολύ. Και σας κύριε Κέρκοπ. Και σας κύριε Γιακολίνο. Θα πρέπει όντως να επεξεργαστούμε αυτή την υπόθεση της ελεύθερης διακίνησης των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Γιακολίνο μας μίλησε για την αρχή της κοινωτικής αλληλεγγύης, δηλαδή να μην υπάρχουν θεσμένες διακρίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι να αισθάνονται ίσοι προς τους άλλους και επίσης θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Κέρχοβ. ε, όντω θα πρέπει να βαθμιστεί η συνεργασία μεταξύ των εργατών μέλων και έτσι να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα των ε, ξένων, των μεταναστών εργαζομένων και επίση να εξασφαλιστεί το ότι οι αρμόδιε εθνικέ αρχέ θα πρέπει μεταξύ του να συνεργάζονται καλύτερα. Πάρα πολύ θετικά είναι τα, τα μαντάτα ότι θα έχουμε αυτού του είδου την εκστρατεία ενημέρωση για του εργαζόμενου ε, του μεταναστέ από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι απαραίτητο ε, γιατί θα πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Και ελπίζω ότι όταν έρθει η ώρα να αναθεωρηθεί ο οργανισμός 16 του 2008 θα καλυφθούν οι προτάσεις μας. Σας ευχαριστώ όλους και ευελπιστώ ότι θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε καλά. Ευχαριστούμε και την το λέει Και τώρα, όπως σας προείπα, Προβλέπετε να πάνω στο σημείο 5 δηλαδή να γίνει η ψηφοφορία ηλεκτρονική όσον αφορά την ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών. Ειδική έμφαση στους σαρωτές σώματος. Η έγκριση αυτού του σχεδίου εκθέσεως που συνέταξε η κυρία Σαρτζεντίνη. Θέλετε να κάνετε κάποια εισήγηση. Όχι, τα έχουμε πει επαρκώς λέει και Σαντζεντίνη, όμως θέλω να σας πω ότι κάτι άλλαξε τελευταία στιγμή στον κατάλογο για την ψηφοφορία. Πρόκειται για την ε, τροπολογία 19. Στην αρχή είχα πει ε, να καταψηφιστεί, τώρα όμως το άλλαξα, έχω βάλει το σημείο συν, θέλω να επιψηφιστεί. Το μείον έγινε συν στην τροπολογία 19. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση και τώρα συνεχίζουμε για την ψηφοφορία. Αρχίζουμε. Για βεβαιωθείτε ότι έχετε την κάρτα. Αρχίζουμε. Συμβαστική τροπολογία παριθμόν 1. Όχι, α, α, διορθώνει ο πρόεδρος. Α, ποιοι είναι υπέρ. Κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία παριθμόν 1. Έχει χωριστεί σε δύο τμήματα το πρώτο. Ποιοι είναι υπέρ. Καταπίπτει όμως διότι εγκρίθηκε το α, διορθώνει ο πρόεδρος. Όμως πρέπει να ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα. Είναι υπέρ. Δεύτερο τμήμα. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τοπολογία. 5. Α, όχι, όχι, όχι. όχι. Συμπαθάτε με πρόεδρος 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το 9. Ψηφίζουμε. Πέρας. 19-21. Επομένως απορρίπτεται. Εκτός μικροφώνου κύριε Σπικέ. Ψηφίσατε αρνητικά όχι υπέρ. Αν ψηφίσατε υπέρ, έχουμε 20-21. Απορρίπτεται. Όπως πριν, επομένως. Πάμε τώρα στο 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 12. Υπέρ. κατά αποχές νομίζω απορρίπτεται 13 έλεγχος για το 12 ψηφίζουμε 12 πέρασε η 25 17 εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές έλεγχος κάνουμε έλεγχο για το 14 ψηφίζουμε πέρας 24-17 εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα το 17 σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται επίσης 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 και 23 που είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 24 καταπίπτει και το 25 και το 26 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας κάνουμε έλεγχο για το 28. Τώρα ψηφίζουμε. 28. Πέρας. 19-24 απορρίπτεται. 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για το 29. Ψηφίζουμε. Πέρας. 22-20 εγκρίνεται. Ε, συμβιβαστική Β υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα έχουμε κάποιες οι οποίες ε, καταπίπτουν μέχρι για την, 35, για το 36 υπέρ, κατά, αποχές, α, απορρίπτεται. 37 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 38 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κόλιο. Δεν έχω την, το κείμενο της μετάφρασης. Και άρα, αφού υπάρχει αυτό το πρόβλημα, δεν θα πρέπει να ψηφιστεί. Άρα το 39 δεν θα ψηφιστεί. Και πάμε στο 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 41. Υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος για το 41. Ψηφίζουμε. Πέρας. 25-18 εγκρίνεται. 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 43. Αποσύρεται. 44. Πέρα. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική γάμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα καταβλήτουν μερικές από τις επόμενες και πάμε στο 51. 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική δέλτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά καταπίπτουν οι επόμενες αρκετές και πάμε στη συμβαστική ε νομίζω. Ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα και μερικές καταπίπτουν και πάμε στο 68. 68 καταπιπτεί. Τότε πάμε στο F, σίγμα ταφ. Υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα καταπίπτουν μερικές και πάμε κατευθείαν στο 78. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω εγκρίνεται. 79. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 80. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 81 υπέρ όχι θα κάνουμε πρώτα έλεγχο για την ψηφορία του 80 Απορρίπτεται 23-19. 81. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 82 κατέπεσε 83 κατά εποχές εγκρίνεται 84 υπέρ κατά ε, εποχές και εγκρίνεται 85 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 86 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για το 86 τώρα ψηφίζουμε για το 86 πέρασε 25-17 εγκρίνεται 87 και 88 έχουν αποσυρθεί και πάμε στο 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται και τώρα το σύνολο του κειμένου όπως τροποποιήθηκε, τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Πέρας. 41-3. Συγχαρητήρια κυρία Σαρτζεντίνη. Και θα πρέπει τώρα να πάμε στο 7, λέει ο Πρόεδρος, το οποίο αφορά την κατάσταση και τη στάση της τρομοκρατίας στην ΕΕ, έκθεση του 2011. Έχουμε και πάλι μια παρουσίαση από πλευράς του Διευθυντή της Ευρωπόλ, του κυρίου Ρομπ Wainwright. Ε, καλώς ορίσατε και πάλι στην Επιτροπή μας. Καθίστε παρακαλώ και ε, ησυχία. Όπως σας είπα, καλωσορίζουμε τον κύριο Rob Wainwright, ε, διευθυντή της Europol, στην Επιτροπή μας για να μας παρουσιάσει την κατάσταση και τις τάσεις της τρομοκρασίας στην ε, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση το 2011, το λεγόμενο TISAT. Θα ακούσουμε την παρουσίασή του και μετά θα ξεκινήσει η συζήτηση. Κύριε Διευθυντά, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι, ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσω τα στοιχεία τα οποία έχετε ε, σήμερα μπροστά σας. Έχετε την παρουσίασή μου για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που βασίζεται εις τα σχόλια των τον των μελών και ε, ορισμένοι άλλοι όπως η Ιντερπολ και άλλοι ε, όπως και θεσμικών οργάνων όπως το Eurojust. Ε, βλέπουμε ότι η τρομοκρατία συνεχίζει να παρουσιάζει πρόβλημα και ε, θα ε, ελπίζω θα το συζητήσουμε και σήμερα το απόγευμα ή στην ακρόαση σχετικά με την αντιτρομοκρατική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταρχής βάσει στατιστικών έχουμε ορισμένες αντενδείξεις όσον αφορά την τρομοκρατική δραστηριότητα δηλαδή δηλαδή έχουν γίνει διάφορες κινήσεις από εθνικιστικές οργανώσεις αλλά η τάση είναι καθοδική σε σχέση με πέρυσι όσον αφορά ε, τις ε, ε, διάφορες, τα διάφορα στοιχεία σχετικά με τις συλλήψεις υπάρχει πάλι μία μείωση ο κίνδυνος είναι αρκετά υψηλός ακόμη λόγω αυξήσεως των απειλών που εκφράζονται από Ισλαμιστικές οργανώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση το τελευταίο έτος και βλέπουμε και ε, ε, μία διαφορετική ε, εμφάνιση γιατί ε, ε, δεν ε, υπάρχει στήριξη αυτής της τρομοκρατικής οργάνωσης και των σχέσεων μεταξύ οργανωμένου εγκλήματος και τρομοκρατίας. Ε, όσον αφορά τις στατιστικές. Ε, το 2010 ε, σκοτώθηκαν και είχαμε και πολλούς τραυματισμούς λόγω των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων που είναι ίδια ρυθμοί όπως και για το 2009. 149 επιθέσεις ήταν, ε, έλαβα χώρα σε εννέα χώρες και οι περισσότερες από αυτές τις επιθέσεις και πάλι έχουν σχέση με ε, ε, τις, τα κινήματα διαχωρισμού στη Γαλλία και στην Ισπανία και μειώθηκαν κατά 50% σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό το 2009 οι ε, οι ε, απειλές αυξήθηκαν το 2010 σε σχέση με το 2009 και όσον αφορά τις ε, δραστηριότητες ε, τρομοκρατών διαπιστώσαμε όπως σας είπαμε ε, υψημένες ενδείξεις ισλαμιστικών κινήσεων το 2010 στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε τρεις ισλαμιστικές επιθέσεις δύο στη Σουηδία, μία στη Δανία με ελάχιστα ζημίες αλλά μία τουλάχιστον με σημαντικά θύματα και αυτό αποτελεί μία μικρή αύξηση. Συγχρόνως όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη και την αποτυχημένη απόπειρα της Αλκάιντα τον Νοέμβριο 2010 εις την ε, ε, Αραβική Χερσόνησο ως ένα αεροπλάνο το οποίο κατευθυνόταν προς της, ε, προς το Ενωμένο Βασίλειο έχουν, ε, είχαμε 179 ε, συλλήψεις περισσότερες δηλαδή από ό,τι τον προηγούμενο χρόνο σε σχέση με το θέμα αυτό και οι μισές από αυτές τις συλλήψεις οφείλονται στην προετοιμασία για τέτοιες απόπειρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια αύξηση δηλαδή 10% σε σχέση με πέρυσι και οι πόλεις που ε, συνελήφθησαν έχουν σχέση με τη χρηματοδότηση και την ε, ε, και την, τον προσιλητισμό τρομοκρατών. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπήρξε μεγαλύτερη ένταση προετοιμασία όσον αφορά δε τις Ισλαμιστικές ε, τρομοκρατικές οργανώσεις ο κίνδυνος είναι μεγάλος στην Ευρώπη και έχουν αυξήσει οι απειλές κατά τους τελευταίους 12 μήνες βλέπουμε και ε, περισσότερη ποικιλία δράσεων από τους Ισλαμιστές υπάρχουν οργανωμένες ομάδες αλλά και και μεμονωμένα άτομα τα οποία κινούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο έλεγχος και η κατεύθυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μέσα έχει μειωθεί ε, κατόπιν των ε, σημαντικών συλλήψεων οι οποίες μας έδειξαν ότι επρόκειτο ή για μεμονωμένους δράστες ή για μικρές μονάδες ε, τρομοκρατών. Οι δραστηριότητες των τρομοκρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, επηρεάζεται και από την, ε, το διεθνές περιβάλλον και το 2010 είχαμε τρομοκρατικές ενέργειες κατόπιν της κατάστασης στη Βόρειο Αφρική. Όσον αφορά την τζιχάντ, την κατάσταση στον, στο Αφγανιστάν, στο Πακιστάν και στο Ιράκ ε, θεωρούμε ότι υπάρχει κίνδυνος να επανέλθουν οι κινήσεις αυτές προς την Ευρώπη διότι το Μάιο 2010 διελήθη στη Γαλλία μία, ένα σημαντικό δίκτυο τρομοκρατών το οποίο ε, είχε προσιλητήσει ε, νέα τρομοκράτες οι οποίοι είχαν εγκαταλείψει τη Γαλλία μεταξύ του 2009 και 2010 για να, ε, ε, ε, για να μεταβούν στο Αφγανιστάν και είχαν προσιλητιστεί στην επιστροφή τους στη Γαλλία διότι βρήκαμε σημαντικά στοιχεία και οι γαλλικές αρχές μπόρεσαν να ξεγελάσουν τις προσπάθειές τους να προβούν σε αυτές τις επιθέσεις πέραν ε, ε, βεβαίως υπάρχουν διάφορα θύματα αλλά πέραν του Πακιστάν, του Αφγανιστάν και του Ιράκ μπορεί να υπάρξουν εθελοντές οι οποίοι προσιλητίζονται και για άλλες κινήσεις. Πέραν των δραστηριοτήτων αυτών, όπως σας είπα, οι περισσότερες επιθέσεις μειώθηκαν το 2010, αλλά διαχωριστικές επιθέσεις ε, σημειώθηκαν στην Γαλλία και στην ε, Ισπανία. Ε, μία δολοφονία υπήρξε από την ΕΤΑ στη Γαλλία και ε, μπορέσαμε να προβούμε σε περισσότερες συλλήψεις. Ορισμένες ορμοκρατικές οργανώσεις όπως η ΕΤΑ και το ε, ΠΚΚ βασίζονται σε εκβιασμούς για να χρηματοδοτήσουν τη δράση τους εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως ε, σε σχέση με επαφές μεταξύ ΕΤΑ και στην Κολομβία διαπιστώσαμε τέτοιες διασυνδέσεις. Υπάρχουν πολλές επιθέσεις στην Ευρώπη και η αύξηση της βίας οδήγησε σε έξι θανατηφόρα επεισόδια το 2010 και συλλάβαμε 34 άτομα που είναι μία αύξηση σε σχέση με πέρυσι. Ορισμένες επιθέσεις οφείλονται σε διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ Ισπανίας, Ιταλίας και Ελλάδος και βλέπουμε ότι υπάρχουν κοινοί στόχοι οι οποίοι επιλέγονται σε διάφορες πόλεις από διάφορες ομάδες σε αλληλεγγύη προς φυλακισμένους συναδέλφους και όπως ξέρετε ε, υπάρχουν υπάρχουν επιθέσεις τα ε, κατά ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και ευρωπαίων πολιτικών σε συντονισμένες ενέργειες από αυτές τις τρομοκρατικές ομάδες. Το 2010 αυτή, αυτά τα αναρχικά αριστερά κινήματα βασιστήκαν στην οικονομική ύφουση η οποία οδήγησε όχι μόνο σε πολιτική ύφεση αλλά οι ορισμένες χώρες στην πρόκληση και ακροδεξιών και ακροαριστερών δραστηριοτήτων. Δεν υπήρξε κάποιο σημαντικό γεγονός το 2010. Βλέπουμε όμως ότι οι εξτραμιστικές οργανώσεις είναι πιο επαγγελματικές, καλύτερα οργανωμένες, ε, ε, χρησιμοποιούν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα για προσιλητισμό και ε, για εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους προσπαθώντας ιδίως να προσελκύσουν νέους σε σχέση με αυτό το οποίο ονομάζουμε εξτρεμισμό επί ενός μόνου θέματος είδαμε ότι υπήρξαν και περιβαλλοντολογικές δραστηριότητες το 2010 πάλι βάσει δικτύων χρησιμοποιώντας τα, τους σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας για να στηρίξουν τις άμεσες ε, ενέργειες και υπήρξε μία προσπάθεια προσπάθεια μετακίνηση των δράσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο προς άλλα μέρη της Ευρώπης, ιδίως ε, το 2010. Εν τω μεταξύ, ε, ορισμένοι αναρχικοί που προστατεύουν τα δικαιώματα των ζώων ε, και εξτρεμιστές είχαν κοινούς στόχους. Ε, πέραν αυτού υπάρχουν και άλλα κοινά θέματα και όπως σας είπα στην αρχή της παρουσίασής μου υπάρχει πολύ ε, κρίσιμη ε, κρίσιμο συντονισμό ιδίως όσον αφορά τον προσιλητισμό και τα μέσα επικοινωνίας και ε, άλλο που μας ανησυχεί είναι ο συνδυασμός μεταξύ τρομοκρατίας και οργανωμένου εγκλήματος διότι πρόκειται ε, για διαφορετικά θέματα τα οποία προσπαθούν να βασιστούν σε ορισμένα προγράμματα ε, και σε κοινά σχέδια βλέπουμε ότι ε, βασίζονται στο εμπόριο λευκής σαρκός ναρκωτικών, ε, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και εκβιασμούς για να χρηματοδοτήσουν αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες και ορισμένες ομάδες όπως το ΠΚΚ επίσης επιδίδονται στο εμπόριο λευκής σαρκός για και ανθρώπων για να χρηματοδοτήσουν τις δράσεις τους και στην Αυστική διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν ενέργειες σε σχέση με ε, την τρομοκρατία στην περιοχή του Σαχέλ ιδίως ε, αυτή την ε, εποχή ασταθείας στη Βόρειο Αφρική υπάρχει μία νέα δραστηριότητα που αναπτύσσεται και ε, συγκεντρώνονται άτομα και οπλισμοί για κινήσεις εναντίον της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Όσον αφορά αυτόν τον απολογισμό του 2010 πιστεύω ότι πολλοί ε, συλλήφθησαν πριν την προετοιμασία ε, των επιθέσεων πιστεύουμε όμως ότι υπάρχει ακόμη μεγάλος κίνδυνος και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να επενέσω την εργασία της αστυνομίας και άλλων ε, αποτρεπτικών οργανώσεων που πρόλαβαν τέτοιου είδους ε, ε, δράσεις και υποβάλλω την έκθεσή μου στην ομάδα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αρκετοί έχουν ζητήσει τον λόγο. Έχω στον καταλογό μου ο κύριος Δίας Ντεμέρας πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε ε, και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, Διευθυντή της ε, Europol για όλα αυτά που μας είπε για την τρομοκρατία. Έχω να κάνω κάποια σχόλια για αρκετά σημαντικά θέματα. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να λάβουμε υπόψη μας ότι η απειλή είναι μόνιμη και η απειλή δεν είναι κάτι που πρέπει να την αγνοήσουμε γιατί υφίσταται αυτή η απειλή όπως πολύ πρόσφατα επισήμανε και η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας. Είναι λοιπόν σημαντικό να επισημάνουμε τη σημασία που έχει αυτή η απειλή σε επίπεδο διαδικτύου. Πόσο σημαντικό είναι το διαδίκτυο. Ε, όσον αφορά στον προσιλητισμό, στη στρατολόγηση ε, και στην προπαγάνδα που ασκείται. Ε, υπάρχουν κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι έχει και άμεση σχέση με την χαρτογράφηση της τρομοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί διώχθηκαν στην Ισπανία. Διαπιστώθηκε λοιπόν αυτή η τάση από το 2009 και μέχρι σήμερα. Ε, πρόκειται για, τον ε, αυτονομιστικό, για την αυτονομιστική τρομοκρατία της ε, ΕΤΑ. Βέβαια έχει μειωθεί ο αριθμός των κατηγορουμένων, όμως ε, στην Ισπανία εξακολουθεί να υπάρχει ακόμα μεγάλος αριθμός ε, επιθέσεων. Έχουμε και αποτυχημένες απόπειρες εκ μέρους ε, των Ισλαμιστών της αριστεράς. Η Γαλλία είναι στη δεύτερη θέση και η Ιταλία στην τρίτη όσον αφορά κυρίως την τρομοκρατία της αριστεράς. Όσον αφορά τον Ισλαμικό, την Ισλαμική τρομοκρατία, στο Βέλγιο και στην Δανία είχαμε σε νέα περιπτώσεις καταδίκες. Ε, πρόσκληση της Europol να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση της ε, τρομοκρατίας. Ε, ως προς αυτό, σήμερα το απόγευμα, όπως ξέρετε, θα έχουμε και μια σχετική ακρόαση για το θέμα αυτό. Πριν κλείσω, θέλω να πω κάτι το οποίο κατά την άποψή μου προσθεθεί στην έκθεση της Σοφή. Οι διαπραγματεύσεις με τους τρομοκράτες πέρα από διαδικαστικής φύσεως θέματα όπως η παράδοση των όπλων ή οι εγκλισμοί σε φυλακές. Τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις ενισχύουν από πλευράς τακτικής τους τρομοκράτες και οι διαπραγματεύσεις αυτές τελικά οδηγούν στην αποδυνάμωση της ασφάλειας και επίσης και στην ε, μεγαλύτερη συμπερίληψη της ε, πολιτικής. Θέλω λοιπόν να πω, κλείνοντας, ότι η διεθνής ε, συνεργασία είναι απολύτως απαραίτητη και το PNR, ο αριθμός των επιβατών, είναι επίσης απαραίτητο. Με αυτές λοιπόν τις παρατηρήσεις ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, τη συνάδελφο για, τις, ε, για την εισήγησή της. Κοιτάξτε, δεν έχω επιβάλει μέγιστο χρόνο ομιλίας, αλλά σας παρακαλώ να είσαστε σύντομοι έτσι ώστε να έχει και κατόπιν ο διευθυντής της Europol αρκετό χρόνο για να απαντήσει. Η κυρία Γκόμες, επόμενη ομιλήτρια. Μικρόφωνο παρακαλώ. είπατε ότι ε, υπάρχει μία διασύνδεση στον τομέα της χρηματοδοτήσετε. Ε, παρακαλώ ελάτε από εδώ γιατί ε, αυτό το μικρόφωνο λειτουργεί ενώ το άλλο δεν λειτουργεί. Είπατε ότι υπάρχει άμεση διασύνδεση, ευξημένη ε, διασύνδεση μεταξύ τρομοκρατίας και οργανωμένου εγκλήματος στο θέμα της χρηματοδότησης. Βέβαια οι ε, υπερπόντιες εταιρείες είναι πολύ σημαντικές σε αυτό το τομέα, οι offshore δηλαδή. Ε, και συμφωνείτε με την άποψη των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων επί του θέματος για έλεγχο των υπερποντίων εταιριών για να μην μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή την αυξανόμενη διασύνδεση τρομοκρατίας και οργανωμένου εγκλήματος και έχετε τεκμηριώσει ε, τέτοιες ε, κινήσεις. Επίσης θα ήθελα να αναφέρω ε, ότι τονίσατε την τάση η οποία υπάρχει στο Σαχέλ και ιδίω τις σχέσεις μεταξύ ε, <clears throat> των ε, εμπόρων ναρκωτικών ε, στη, στη Νότιο Αμερική με ε, ορισμένες ε, κινήσεις σε διάφορες χώρες. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω όσον αφορά τις έκτακτες παραδόσεις υπάρχουν πάρα πολλές αδυναμίες εις τα αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής Ενώσεως ιδίως εις την ε, Ιβηρική Χερσόνησο όπου επικεντρώνονται αυτές οι τρομοκρατικές ε, δραστηριότητες. Γίνεται καμιά κίνηση για να βελτιωθεί ε, αυτό το σύστημα. Ο κύριος Κύρκοφ, σας ευχαριστώ κύριε Γουίνραιτ πάρα πολύ για την έκθεσή σας. Τη σχεδιάστε, την παρουσιάσετε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως η έκθεση αυτή είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα για αυτά που δεν περιλαμβάνει από αυτά που περιλαμβάνει. Και η επιτυχία που σημείωσαν οι άντρε σα ε, στις επιχειρήσεις τους ξέρουμε πολύ καλά ε, ότι είχαν επιτυχίες, ε, δεν τις ξέρουμε με λεπτομέρειες, αλλά υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι υπάρχουν επιτυχίες στη δουλειά που κάνατε και σας είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό και σε εσά και στους συναδέλφους σας. Σύντομα λοιπόν θα ρωτήσω η ροή ανθρώπων από τη Βόρεια Αφρική αυτή τη στιγμή και η συμμετοχή των δυνάμεων ε, των κρατών μελών μέσα από το ΝΑΤΟ. Αναφέρομαι στην επίθεση στη Λιβύη. Αυτό πώς επηρεάζει αυτή τη στιγμή τη σκέψη σας και την στρατηγική στρατηγική ασφάλεια που εφαρμόζεται με τον τρόπο αυτό αυξάνεται ή όχι ο κίνδυνος της ε, τρομοκρατίας και ως εισηγητής ε, στη νέα συμφωνία ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το PNR και επίσης και σε σχέση με την οδηγία για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, αυτά τα δύο θέματα πώς πιστεύετε ότι θα βελτιώσουν τη δουλειά σας κατά την επόμενη, αυτήν και την επόμενη χρονιά. Ο κύριος Άλμπρεχτ. Ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ και τον ε, κύριο Βάινράιτ για την ε, παρουσίασή του. Ακούσαμε την έκθεσή σας ε, και εκείνο που με απασχολεί είναι το εξής. Είναι αρκετά δύσκολο να παρακολουθήσει κανείς τη συζήτηση ε, για τον, ε, την τρομοκρατία, γιατί δεν υπάρχει ορισμός της ε, τρομοκρατίας στην έκθεσή σας. Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι αυτό είναι κάτι για το οποίο πρέπει να συζητήσουμε περισσότερο, κυρίως σε σχέση με τις τρομοκρατικές ενέργειες τις οποίες αναφέρεστε. Διότι κατά τη δική μου άποψη πάρα πολλά από αυτά που αναφέρετε στην έκθεσή σας δεν θα έλεγα ότι είναι φυσιολογικά, σε εισαγωγικά, αλλά αν θέλετε πρόκειται για καθαρά οργανωμένο έγκλημα, επικίνδυνο έγκλημα, αλλά δεν πρόκειται για τρομοκρατία. Και αν θέλετε να αξιολογήσουμε την τρομοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχουμε σαφή ορισμό ε, για να ξέρουμε τι μιλάμε. Αυτό είναι απαραίτητο, διότι κατά την άποψή μου μετακινούμεθα όλο και περισσότερο στο να συγκεντρώνουμε εγκλήματα διαφορετικών μορφών μέσα σε, αυτό, σε αυτή τη μεγάλη χωάνη της ε, τρομοκρατίας όπου μπορούμε να πούμε, κάποια στιγμή θα πούμε ότι υπάρχει ακόμα και ε, αθλητική τρομοκρατία, το λέω έτσι καθ' υπερβολή. Αλλά εν πάση περιπτώσει οποιασδήποτε μορφή σε έγκλημα πολύ εύκολα μπορεί να αποδοθεί στην, σε τρομοκρατική δραστηριότητα. Εκείνο που μας ενδιαφέρει όμως είναι να εστιάσουμε την προσοχή μας σε ουσιαστικές ε, απειλές ε, που βεβαίως και υπάρχουν. Πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα. Νομίζω όμως ότι θα ήμασταν περισσότερο αποτελεσματικοί αν είχαμε ένα σαφέστερο ορισμό της ε, τρομοκρατίας. Ο κύριος Πίρκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για την έκθεση γιατί παρουσίασε με μεγάλη σαφήνεια ότι η απειλή εξακολουθεί να είναι εξίσου έντονη. Ω εκ τούτου και αρμόδιες αρχές καλούνται να προσαρμόσουν την στρατηγική τους. Εγώ έχω τέσσερα ερωτήματα. Το πρώτο είναι το εξή. Αυτή τη στιγμή συζητάμε για την ε, χρήση των σαρωτών ασφαλείας, των σκάνερ και εσείς ε, πώς ε, το συνδέεται αυτό με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ε, τρομοκρατίας. Δεύτερη ερώτηση. Αναφερθήκατε στην όλο και μεγαλύτερη συνεργασία, διασυνοριακή συνεργασία τρομοκρατών. Και ρωτώ, εντωμεταξύ τα δεδομένα που δίνουν τα κράτη-μέλη αρκούν έτσι ώστε η Europol να μπορεί να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Τρίτο ερώτημα αφορά στις όλο και περισσότερες συλλήψεις, πολύ καλές αυτές, αλλά αυτές τις συλλήψεις σε ποια ακριβώς μέτρα τις ανάγεται. Και τελευταία μου ερώτηση είναι η εξής. Αναφερθήκατε σε πηγές χρηματοδότησης τρομοκρατικών δραστηριοτήτων και ερωτώ. Έχετε κάποια εμπειρία, γνωρίζετε μήπως ε, για το ε, εμπόριο, τη διακίνηση, την με διακίνηση ανθρώπων. Ε, θεωρείτε ότι αυτή είναι πραγματικά μια πηγή χρηματοδότησης για την τρομοκρατία στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Χαιρόμαστε ιδιαίτερο που επανήλθατε σε αυτό το κοινοβούλιο. Έχω οκτώ ονόματα εδώ. Έχουμε μισή ώρα ακόμη. Μέχρι στιγμής ήσασταν πολύ πειθαρχισμένοι. Αν είσαστε ε, έτσι θα έχει ο καθένας δύο λεφτά και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε έτσι. Κύριος Κροτσέτα. Έχω να υποβάλω κάποιες ερωτήσεις. Παραδείγματος χάρη, όσον αφορά στην Ιταλία, θα μιλήσω ε, για την Ιταλία, αλλά το πρόβλημα υπάρχει και σε άλλες χώρες. Στην Ιταλία, ας πούμε, γίνεται λόγος για τέσσερις Ισλαμικές επιθέσεις, έξι αυτονομιστικές, οκτώ επιθέσεις ε, ε, εξ αριστεράς και κάποιες άλλες επίσης από την δεξιά. Εγώ ζω στην Ιταλία και δεν είχα, λάβει, δεν είχα πάρει είδηση από αυτές τις απόπειρες. Θα ήθελα να ξέρω το επίπεδο στο οποίο κατατάσσεται τις ε, επιθέσεις αυτές. Δηλαδή, τι είναι εκείνο το οποίο οδηγεί στο να χαρακτηριστεί μία επίθεση ως τρομοκρατική επίθεση. Παραδείγματος χάρη, ε, το γεγονός ότι πέταξαν αυτό το αγαλματάκι ε, στο πρόσωπο του Μπελουσκόνη αυτό ήταν τρομοκρατική επίθεση ή όχι. Ε, σίγουρα ήταν κάτι το ε, καταδικαστέο. Αυτό όμως ήταν μια πράξη παράφρονα και δεν ήταν αποτέλεσμα μιας στρατηγικής. Άρα δηλαδή μια πράξη για να χαρακτηριστεί τρομοκρατική θα πρέπει να έχει προκύψει μετά από κάποια συγκεκριμένη στρατηγική. Άλλο ερώτημα. Το οργανωμένο έγκλημα. Υπάρχουν και τρεμοκρατικές ενέργειες που χαρακτηρίζονται ως τρομοκρατικές. Υπάρχουν λοιπόν εγκληματικές πράξεις, το, οργανω... το έγκλημα είναι οργανωμένο σε ολόκληρη την Ευρώπη και αναμφίβολα έχει διαπράξει πολλές περισσότερες ε, επιθέσεις. Αν δημοσιευτούν τα στοιχεία πραγματικά θα τρομάξετε. Ανταυτού όμως ε, δεν έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία, δεν αναφέρονται στοιχεία αυτά στις εκθέσεις. Μερικές φορές ε, μιλάμε για βόμβες που ανατινάσσονται, που εκρήγνονται. Μετά μιλάμε για δημάρχους που δολοφονούνται, πολιτικούς, δικηγόρους, δημοσιογράφους, δικαστές. Αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλές χώρες. Ακόμα λοιπόν ε, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία για όλα αυτά. Και τελευταία μου ερώτηση. Η Μεγάλη Βρετανία. Γιατί η Μεγάλη Βρετανία δεν μπορεί, δεν έχει κατορθώσει να χαρακτηρίσει τις επιθέσεις που έχουν λάβει χώρα στη δική της ε, την επικράτεια ως τρομοκρατικές ή όχι. Ε, νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει ένας σαφής ορισμός για την τρομοκρατία έτσι ώστε να αποφύγουμε η όλη προσέγγιση να είναι καθαρά ιδεολογική και να αποφύγουμε η τρομοκρατία να γίνει το επίκαιρο θέμα ενώ οι μαφίες συγκεκριμένου να διαπράττουν δολοφονικές ενέργειες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο κύριος Μπουσουτήλ. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Wayne Ράιτ για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίασή του και για την εργασία την οποία κάνει. Ένα από τα θέματα τα οποία διαφαίνονται ε, και προσέλκυσε την προσοχή μου είναι η μελλοντική ροή μεταναστών από τη Βόρειο Αφρική που μπορεί να επηρεάσει την κατάσταση ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και είπατε ότι άτομα με τρομοκρατικούς στόχους μπορεί Δηλαδή να παρισφρήσουν στους ε, μετανάστες αυτούς και ε, θεωρώ ότι αυτό είναι ε, πάρα πολύ επικίνδυνη δήλωση βάσει τίνο στοιχείου το, λέτε ε, τι κάνει η Ευρωπόλ για να αντιταχθεί σε αυτές τις προσπάθειες και θα ήθελα να ξέρω αν έχετε στείλει μία απαστολή ή ορισμένους σε χώρους όπως η Μάλτα και η Ιταλία όπου υπάρχει μία αύξηση αυτών των προσφύγων ο κύριος Παπα-Νικολάου. Mr. Thank you. Κύριε Βέινρατ, ε, σας ευχαριστώ και πάλι για αυτή την παρουσίαση. Όλα αυτά τα οποία μας είπατε είναι πολύ σημαντικά. Έχω την εξή ερώτηση. Αναφέρατε τον ευξημένο συντονισμό μεταξύ τρομοκρατών σε διάφορα κράτη-μέλη. Επίσης αναφέρατε το διαδίκτυο σαν διευκολυντή αυτών ε, των ε, τάσεων. Διαπιστώνω ότι έχουμε ε, συλλήψεις τρομοκρατών μόνο σε 15 από τις 27 χώρες. Αυτό οφείλεται γιατί δεν έχετε πληροφορίες από τα άλλα 12 κράτη-μέλη ή έχουμε άλλα προβλήματα για τα οποία θα πρέπει να ενημερωθούμε. Ο κύριος Μωράης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο Wainwright της ομάδας μας ε, για την εργασία, ευχαριστώ το, εκ της ομάδας μας τον κύριο για την εργασία που κάνει. Η έκθεση αυτή είναι πολύ σημαντική και βλέπω ότι ο κύριος Άλμπερεχτ ρώτησε ε, για τον ορισμό της τρομοκρασίας πράγμα που ρώτησε και ο κύριος Κροτσέτα ξέρω ότι στο έγγραφο αυτό υπάρχει ένας τέτοιος ορισμός θα ήθελα όμως εδώ να περιοριστώ σε ένα ερώτημα λόγω του χρόνου ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχει μια στρατηγική εσωτερικής ασφαλείας σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα ε, θα ήθελα λοιπόν να ξέρω ποια είναι η μεγαλύτερη απειλή κατά την αξιολόγηση της Ευρωπόλ και πώς εσείς πιστεύετε ότι οι πόροι σας χρησιμοποιούνται για αντιτρομοκρατικές ενέργειες διότι υπήρξε μία επίσημη, μία επίσημη επίθεση κατά αυτών των δράσεων τις οποίες θεωρώ όρισαν σαν σφατάλι και αυτό έγινε στι Ηνωμένε Πολιτείε. Οπότε λαμβανομένων υπόψη του τι κάνει το ΝΑΤΟ στη Βόρειο Αφρική μήπως θα έπρεπε να παρακολουθήσουμε και να εστιαστούμε πολύ συγκεκριμένοι και να αξιολογήσουμε ακριβώς πού είναι οι απειλές μας πριν αρχίσουμε να βλέπουμε τις επικεφαλίδες της εφημερίδας Πώ Πώς δηλαδή πιστεύετε ότι μπορούμε να συνδυάσουμε τους δύο στόχους μας, ο κύριος Σταβάρες. <laughs> Πρέπει να σας πω σαν πράσινη ότι περάσαμε μέσα από την αίθουσα και ε, απενεργοποιήσαμε τα, τα τα μικρόφωνα. Σαν ε, πράσινος λοιπόν, εφόσον βλέπω ότι μόνο αυτά τα μικρόφωνα λειτουργούν, θα ήθελα να σας πω ότι καταρχήν βεβαίως δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί πλήρης και απόλυτη ασφάλεια, αλλά κάτι δεν πάει καλά στον τρόπο με τον οποίο πολλές φορές υπολογίζουμε το επίπεδο της απειλής που φαίνεται ε, πιο ήπιος και λέτε έχουμε λιγότερες ε, τέτοιες επιθέσεις ενώ στην πραγματικότητα η απειλή είναι πιο σοβαρή πράγμα το οποίο μας δείχνει ότι δεν είναι γραμμική η απειλή αλλά πολύ πιο ασαφής οπότε ε, υπάρχουν διάφορες ε, δυνατότητες και ε, ε, φαίνεται πιο απλή η κατάσταση από ό,τι όντως είναι. Γι' αυτό και πρέπει πολιτικά να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό και that they have ε, reasons for recruitment. This is, in my sense, addressing it politically διότι η καταστολή ε, επιτυχάνει, όχι όμως πάντοτε, ορισμένες φορές είναι αντιπαραγωγική και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε προσέλκυση ε, τρομοκρατών, ε, οπότε ορισμένες φορές καλό θα ήταν να κινούμαστε έξυπνα ως προς το πώς προχωρούμε στο τομέα αυτό διότι ε, πρέπει να μην, ε, να μην κινούμεθα κατά τρόπον ο οποίος είναι εις βάρος των πολιτών και αυξάνει και την προσέλκυση τρομοκρατών. Ε, είναι όμως και θέμα χρηματικό. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δυνατότητα να αμφισβητήσει κανείς τα όρια χρηματοδότησης διότι δεν έχουμε για κανέναν τομέα τεράστιες δυνατότητες χρηματοδότησης ούτε για την εκπαίδευση. Πολλές φορές λοιπόν η καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι δαπανηρή. Μήπως δαπανούμε υπερβολικά για αυτό που επιτυχάνουμε. Ευχαριστώ. Ε, ε, σωστά όμως αναφερθήκατε και στο θέμα του κόσμου, Ο κύριος Μίλντερ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Βέιν Έχω μία απλή ερώτηση να σας υποβάλω. Αν ρίξετε μια ματιά στο πώς έχει η νομοθετική κατάσταση στην Ευρώπη, τι λέτε κύριε Wainwright, είναι επαρκής η νομοθεσία ή θα μας προτείνετε σε εμά και στην Επιτροπή να θεσπίσουμε και άλλα μέτρα. Δηλαδή, σας διευκολύνει όχι στο έργο σας η κείμενη νομοθεσία. Ευχαριστώ πολύ. Και νομίζω ότι αυτή η ερώτηση αφορά και την έκθεση. Τρίτη ερώτηση από πλευρά δική μου, ή μάλλον έχω μία ερώτηση και μία παρατήρηση. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη από αυτή την έκθεση. Ε, νομίζω τα πράγματα πάνε καλύτερα και επομένω έτσι θα ενθαρρυνθούν τα κράτη-μέλη να δίνουν περισσότερε πληροφορίε, γιατί βεβαίω ε, ε, από τι πληροφορίε που μας δίνουν εξαρτάται το τι κάνουμε επομένως ε, καλά πάμε και θα βελτιωθούμε με την πάροδο του χρόνου Τώρα βέβαια το θέμα είναι τι κάνει η Επιτροπή και το Συμβούλιο και όχι εσείς κύριε Wainwright. Εάν κανείς ετήσια κάνει έναν απολογισμό εξετάσει την απειλή και την ε, δρασή μας για να μπορέσουμε πέραν της θεωρητορίας έκθεσης που έχουμε αυτή την εικόνα των τάσεων να δούμε και αυτή είναι η ερώτησή μου σε σχέση με αυτά που είπε ο Γιάνν Άλμπρεχτ και άλλοι όσον αφορά τον ορισμό της τρομοκρατίας γιατί πραγματικά θεωρώ ότι στην πράξη όλο ένα και διευρύνεται ο ορισμός. Για να δούμε ας πούμε. Την ε, σύγκρουση μιας ομάδας αστερών και μιας δεξιών και ε, να έχουμε κάποιο μαχαίρωμα κατά τη ε, συμπλοκή. Αυτό τι είναι, έγκλημα ή τρομοκρατική πράξη. Μια ανθρωποκτονία. Γιατί τώρα αυτό το ονομάζουν τρομοκρατική επίθεση. Επομένως, μέχρι που φτάνει ο ορισμός, δεν θα έπρεπε να χτυπάει την εθνική ασφάλεια και όχι την ατομική ασφάλεια η τρομοκρατία. Όσο για να θέλουμε να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή. Πολλές φορές λέμε ότι πρόκειται για φαινόμενο το οποίο πλήσει γενικότερα την κοινωνία. Και θυμάμαι κάτι που είχε γίνει στις κάτω χώρες πριν από ένα χρόνο. Είχαμε μια διαδήλωση, μάλλον συγκέντρωση χιλιάδων, χιλιάδων λαού. Υπήρχε κάποιο είδου ε, επίσημη εκδήλωση, ήταν, ήρθε και η βασίλισσα, όλοι ήταν ίσχυοι και μόνο ένας, μόνο ένας, ένας μόνο αποδοκίμασε, αποδοκίμασε την ε, βασίλισσα και και έγινε τόσο πανικός που 65 πρόσωπα τραυματίστηκαν. Συνελήφθη αυτός μόνο και μόνο γιατί απεδοκίμασε. Όλη η κοινωνία μας θεωρήσε ότι πάρει εφίσταται επίθεση. Είχαμε έκτακτα δελτία ειδήσεων κλπ. Επομένως είχαμε αντίκτυπο πάρα πολύ σημαντικό. Όμως η επίθεση ήταν μόνο μια κραυγή αποδοκιμασίας. Άρα Πού είναι τα όρια μεταξύ εγκληματικής πράξης και τρομοκρατικής πράξης. Ίσως θα πρέπει να είμαστε πιο επιφυλακτικοί. Αυτές είναι όλες οι ερωτήσεις των συναδέλφων και ελπίζω ότι μπορείτε να τις απαντήσετε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Αντί για μία-μία θα προσπαθήσω να καλύψω ομαδικά τις ε, παρατηρήσεις για την Βόρεια Αφρική. Προβληματίζονται και τα κρατημέλη και η Europol όσον αφορά το κατά πόσον θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε την δημοσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο βαθμό που έχουμε οποιαδήποτε κίνηση στην περιοχή θα μπορούσαν κάποιοι ακραίοι να εκμεταλλευτούν για να στρατολογήσουν πρόσωπα. Το θέμα είναι τι γίνεται με το πολιτικό κενό. Πώς μπορεί το πολιτικό κενό να έρθει από κάποιους που έχουν διαφορετικό πρόγραμμα ο καθένας. Ε, επίσης, όσον αφορά τον βαθμό που η αστάθεια οδήγησε σε μείωση των ικανοτήτων δράσης της αστυνομίας και διοικητικών αρχών. Οπότε και τώρα έχουμε εγκληματικέ και τρομοκρατικέ δραστηριότητε παρόν παρατηρητέ από την αστυνομία. Επίση, τι γίνεται όσον αφορά την ροή μεταναστών από, την, ε, από τι χώρε αυτέ προ την Νότια Ευρώπη. Έχουμε τώρα, έχουν τώρα μόνο την ευκαιρία τρομοκράτε να μετακινούν του ανθρώπου του, αλλά και τρομοκρατικό υλικό, εξοπλισμό. Μέχρι σήμερα πάντως δεν έχουμε στοιχεία για το ότι οι τρομοκρατικέ οργανώσει κάνουν κάτι τέτοιο. Όμω, είναι λογικό να σκεφτεί κανεί κάτι τέτοιο. Παντώ όσον αφορά ε, εγκληματικέ οργανώσει, ναι, το κάνουν αυτό τώρα. Περνάνε ανθρώπου του ε, ε, οι μαφίες από τη μία όχθη της Μεσογείου στην άλλη. Τώρα για τον κύριο Μπουσούδη συγκεκριμένη ερώτηση όσον αφορά την επιχειρησιακή ομάδα της ε, Europol που δύο λεπτά ε, ε, έχουν πάει στην Λαμπεντούσα και επίσης στην πυροτική Ιταλία η Frontex και οι Ιταλικές αρχές προσπαθούν να ζυγίσουν τις πληροφορίες και επίσης γίνεται και κάποια ενημέρωση από πλευράς όσων φτάνουν εκεί. Άρα προσπαθούμε να δούμε σε ποιο βαθμό το οργανωμένο έγκλημα έχει εμπλακεί σε αυτή την κατάσταση. Προς το παρόν, επομένως, δεν υπάρχουν τα ίδια στοιχεία για τρομοκράτες όπως υπάρχουν για τους ε, εγκληματίες. Τώρα, όσον αφορά την υπόλοιπη Αφρική, μας προβληματίζει αυτό το οποίο είπαμε προηγουμένως, ότι Υπάρχουν σχέσεις μεταξύ διεθνών κυκλωμάτων ναρκωτικών και κάποιων στο Σαχέλ που φέρονται ως Ισλαμιστές. Ούτε αμέσως σχέση έχουμε διαπιστώσει να υπάρχει μεταξύ ε, δουλεμπορίας και τρομοκρατίας στην περιοχή. Τώρα όσον αφορά τον ορισμό της τρομοκρατίας. Υπάρχει κάποιος ορισμός και τον χρησιμοποιούμε στην έκθεση ε, και βέβαια θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά το βαθμό στον οποίο καλύπτουμε κάθε τρομοκρατική δραστηριότητα. Όντως, όπως είπατε είναι, το δέχομαι. Και εμείς έχουμε σαν ορισμό αυτόν που ενέκριναν τα κράτη-μέλη. Επομένως θα πρέπει και η έκθεση να ληφθεί υπόψη σε σχέση με τη συνέντευξη αυτή των κρατών μελών. Όντως. Κάνουμε ό,τι λένε τα κράτη-μέλη, δεν είναι δική μας δουλειά. Να, μαντεύουμε τι θεωρεί κάθε κρατός μέλος ε, τρομοκρατία. Ακούμε τι έχουν να πούν τα κράτη-μέλη, συγκεντρώνουμε τα στοιχεία, κάπως όπως αυτή η έκθεση. Ναι, είναι αλήθεια. Η έκθεση βελτιώνεται. Ακόμα υπάρχουν ε, κάποιες αδυναμίες βέβαια. Το ότι ακόμη δεν έχουμε λάβει όλα τα στοιχεία που θέλουμε από τα κράτη-μέλη. Και αυτό μας δείχνει το πόσο δύσκολη υπόθεση είναι η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας στην Ευρώπη. Ας πούμε δεν ξέρουμε τον αριθμό των συλλήψεων, πάντως αυτό είναι ένα μόνο στοιχείο όσον αφορά το επίπεδο στο οποίο κινείται η τρομοκρατία. Όντως δεν έχουμε μια με διαδρομή τώρα. Έχουμε τα ωριά μας όσον αφορά την έκθεση. Ε, περιγράφει την κατάσταση όπως έχει. Αναλύει κάποιε τάσεις. Αλλά δεν ισχύει το ίδιο όπως και με το οργανωμένο έγκλημα. Δεν πρόκειται για έκθεση από τη βάση πλαισιών πληροφοριών. Κάποια στοιχεία τα κράτη-μέλη δεν μας τα δίνουν. Δεν έχουμε πρόσβαση και ούτε μπορούμε να τα δημοσιοποιήσουμε. Και αν τα έχουμε επομένω, αυτά είναι τα όρια τη έκθεση. Πάντω, όντω βελτιώνεται η έκθεση και ιδίω όσον αφορά κάποια ευαίσθητα δεδομένα, νομίζω ότι δείχνουν την κατάσταση που βρισκόμαστε. Για αριστερού, δεξιού, εξτρεμιστέ και τη σχετική δραστηριότητα, ε, αυτά όλα είναι μικρό κομμάτι τη έκθεση γιατί τα περισσότερα αφορούν την ΕΤΑ και ακόμα σε κάποια κράτη-μέλη ε, έχουμε θέματα Ισλαμικής τρομοκρατίας και τα πιο βέστα δεδομένα στην έκθεση δικαιολογούν και εξηγούν το ότι υπάρχει συνεχής απειλή από αυτές τις, αυτά τα κέντρα. Τώρα, η δράση, να μην υπερβάλλουμε, οι περισσότερες ε, οι περισσότερε εγκληματικέ οργανώσει δεν συνεργάζονται με τους τρομοκράτε. Είναι βέβαια κάτι που δεν το αποκλείουμε και ίσω όλο ένα και περισσότερο. Έχουμε τέτοιου είδου διαπλοκή και στην Αφρική έχουμε τέτοιε ενδείξει. Τώρα, όσον αφορά την χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων των ΜΕΝ από του ΔΕ. Έχουμε τώρα πάρα πολλέ ε, ευκαιρίε κάνει να κερδίσουν λεφτά, και να χρηματοδοτηθούν οι τρομοκράτε κυρίως μέσω του διαδικτύου. Επομένως, να πώ προκύπτει η διαπλοκή του, του των μεν με τους δε. Συγκεκριμένη ερώτηση τώρα τη κυρία Γκόμες. Σχετικά με το ε, ξέπλυμα βρώμικου χρήματο ε, και το θέμα των ε, εξωχώριων εταιριών ε, και πολλές άλλες δραστηριότητες ξεπλήματος βρώμικο χρήματος ε, δραστηριότητες που χρησιμοποιούν οι τρομοκρατικέ οργανώσεις. Πρέπει να σας πούμε ότι γι' αυτά αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν έχουμε ε, αρκετέ πληροφορίε. Κάτι άλλο που ετέθη ε, σχετικά με την αντιμετώπιση της τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα. Κατά πόσον δηλαδή υπάρχει συσχετισμό ανάμεσα στα δύο. Ε, και θέλω να σας πω ότι το να μπορεί κανείς να ε, λειτουργήσει στο διαδίκτυο, παραδείγματο χάρη όσον αφορά την αξία ε, της πληροφορίας και την ανταλλαγή πληροφοριών. Βλέπουμε όλο και περισσότερο ότι προκύπτει μια ανάγκη συνεπούς πολιτικής ανάμεσα στην αντιμετώπιση της τρομακρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Και στη Europol εμείς έχουμε καταλήξει ότι θα πρέπει να υπάρχει όλο και μεγαλύτερη συνεργασία όσον αφορά την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τις εθνικές στρατηγικές των κρατών μελών που έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Πρέπει η δουλειά που γίνεται να συνδυαστεί καλύτερα και να ε, συνδυαστούν καλύτερα οι δυνατότητε που υπάρχουν. Για την Europol η τρομοκρατία παραμένει ένα σημαντικό κομμάτι των εργασιών μα, όχι βέβαια το μόνο. Ε, διαθέτουμε 19% των πόρων μα και το 30% το διαθέτουμε ε, στην παράνομη αντιμετώπιση της παράνομη διακίνηση ατόμων. Νομίζω Κάλυψα με ταχύτητα βέβαια τις περισσότερες ερωτήσεις όσον αφορά την εργασία της ε, Europol. Δεν έχω να πω τίποτα συγκεκριμένο για τις αδυναμίες που υπάρχουν στην ε, Ιβυρική Χερσόνησο και στα αεροδρόμια για τους ε, σαρωτές και γι' αυτό δεν μπορώ να προσθέσω τίποτα άλλο. Όσον αφορά τη στρατηγική για το PNR βεβαίω και μια τέτοια στρατηγική ενισχύει την ασφάλεια. Ε, και εμείς ε, προσπαθούμε να μεγιστοποιήσουμε τα ωφέλη που μπορούν να ε, προκύψουν από την ανταλλαγή πληροφοριών. Το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, όπως και άλλες μελλοντικές οδικίες, πράγματι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τη σημαντική αύξηση που διαπιστώνεται στην παράνομη χρήση του διαδικτύου για την στήριξη εγκληματικών ενεργειών και τρομοκρατίας. Η αστυνομία ε, πρέπει να έχει όλο και περισσότερα μέσα κάθε μέρα για να μπορεί να αντιμετωπίσει αυτά τα δύο προβλήματα. Ε, νομίζω ότι κάλυψα τις περισσότερες ερωτήσει, Αν όχι, μπορείτε να έρθετε να με βρείτε κατηδίαν ή μπορείτε και να επανέλθετε. Ο κύριος Μούλντα. Η δική μου η ερώτηση ήταν κατά πόσον η υπάρχουσα νομοθεσία επαρκεί στη Europol ε, για να πραγματοποιήσει το έργο τη ε, ή μήπω επιθυμείτε περισσότερο νομοθετικό έργο. Συγγνώμη κύριε Μούλντα που δεν απάντησα στην ερώτησή σα. Νομίζω ότι σήμερα το απόγευμα στην ανταλλαγή πληροφοριών που θα έχουμε θα εστιάσουμε την προσοχή μα σε αυτό το θέμα. Γιατί πιστεύω ότι ε, έχει σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Ω προ τη Europol θέλω να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δούλεψε πολύ σκληρά στα 10 χρόνια από την 10η Σεπτεμβρίου για να υπάρξει αποτελεσματική νομοθεσία αντιμετώπιση τρομοκρατία. Δεν αποκλείω ότι πρέπει να υπάρχει και άλλο νομοθετικό έργο, αλλά αυτό που ενδιαφέρει είναι αυτή τη στιγμή να εφαρμόζουμε αποτελεσματικότερα την κείμενη νομοθεσία. Ε, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Wainwright. Αν δεν υπάρχουν ε, άλλα σχόλια, από ό,τι βλέπω δεν επιθυμεί κανείς άλλος να σχολιάσει κάτι. Κατόπιν τούτου ε, ολοκληρώσαμε τις εργασίες μας για σήμερα το πρωί και θα επανέλθουμε από τις 3 ε, ε, το μεσημέρι για την ακρόση. Για αυτά τα θέματα Ολοκληρώσαμε όπως σας είπα. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τον κύριο Wainwright για την ε, παρουσία του. Τον ευχαριστούμε για το έγγραφο που μας ε, παρουσίασε ε, και το έγγραφο διατέθηκε σε όλα τα μέλη της Επιτροπής. Εξακολουθούμε να έχουμε βέβαια και λίγο χρόνο ακόμα πριν ξεκινήσουμε και κλεισμένων των θυρών τη συνεδρίαση των συντονιστών. Ευχαριστούμε τον κύριο Ράιτ και στις 11.30 ε, ακριβώς θα αρχίσουμε τη συνεδρίαση των συντονιστών. Σας ευχαριστώ πολύ.